Buonasera a tutti. Cominciamo perché oggi abbiamo eh, i tempi ristretti. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Πρέπει να βιαστούμε. Οι διαθέσιμε γλώσσε είναι στο Info Δεν υπάρχει web streaming, αλλά θα μαγνητοφωνηθεί η συνεδρίαση και όσοι ενδιαφέρεστε μετά να το δείτε μπορείτε να το ζητήσετε. Σας θυμίζω ότι αύριο θα πρέπει να πάρετε τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την ακρόαση των υποψηφίων μελών του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχουμε έξι υποψήφια μέλη του συνεδρίου τα οποία θα ακούσουμε. για κάθε μέλος υποψήφιο έχουμε 30 λεπτά στη διάθεσή μας, γι' αυτό 5 λεπτά θα πάρει η εισαγωγή του υποψηφίου, 5 ή 10 λεπτά για τον εισηγητή που θα θέσει ερωτήσεις, θα υπάρξουν απαντήσεις με τη λογική της επιτραπέζιας αντισφαίρησης και όσοι θέλουν να θέσουν ερωτήσεις πρέπει να το πούνε στον γραμματέα μας τον κύριο Μπράουν. θα είμαι αυστηρός με το θέμα του χρόνου. Όταν ξεπερνάτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας θα σας αφαιρώ το λόγο. Η κυρία Αγιάλα έχει ζητήσει το λόγο. Αγιάλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μόνο από τις διαδικασίες να πω το εξής. Κοιτάξτε, ε, είμαστε στην προπαρασκευαστική ομάδα και πριν από μισή ώρα ακριβώ τότε πήραμε μία επιστολή σε σχέση με τον ε, υποψήφιο που θα πάρει το λόγο. Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι είναι σωστός αυτός ο τρόπος. Ε, ε, κοιτάξτε, χωρίς χρόνο, χωρίς ε, το χρόνο να το εξετάσουμε και να το συζητήσουμε. δεν θέλω, νομίζω δεν πρέπει να την λάβουμε υπόψη αυτή την επιστολή. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη διαδικασία, κυρία Αγιάλα, με το πρόγραμμα έτσι όπως έχει καθοριστεί. Και μετά θα προχωρήσουμε στην αξιολόγησή μας και για την επιστολή στην οποία αναφερθήκατε. Θα ξεκινήσουμε με τον Ούγκρο υποψήφιο, τον κύριο Φαζάκας. Θα δώσω αμέσως το λόγο λοιπόν στον υποψήφιο, ο οποίος έχει πέντε λεπτά στη διάθεσή του για να παρουσιαστεί. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Δεν θα, χρειαστεί νομίζω να επαναλάβω το πόσο ευτυχής είμαι που ξαναβρίσκομαι εδώ σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών με διαφορετική ιδιότητα αυτή τη φορά σαν ο υποψήφιος των Ουγγρικών Αρχών για μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χαίρομαι γιατί γίνεται η συνάντηση αυτή μια 15η Μαρτίου όπου εμείς γιορτάζουμε την Επανάσταση του 1848. Εγώ έχω περάσει εδώ πέντε χρόνια, μία ολόκληρη κοινοβουλευτική περίοδο, έχω κάνει ό,τι μπορούσα, προσπάθησα όπως μπορούσα, ήμουν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών, ήμουν μέλος της Επιτροπής ε, Ελέγχου Προϋπολογισμών όπως είπα και κοσμήτορας κατά δυόμιση χρόνια. Είναι μεγάλη χαρά για μένα λοιπόν που βρίσκομαι εδώ. Προετοιμάστηκα ελπίζω καλά και προσπάθησα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν υπάρχει ανάγκη να συστηθώ λοιπόν περισσότερο, να δώσω κάποιες απαντήσεις σχετικά με το πολιτικό μου παρελθόν ε, δεν έχω να δηλώσω κάποιες πολιτικές δραστηριότητες παρούσες σε ισχύ, δεν έχω να δηλώσω επίσης κάποιες οικονομικές δραστηριότητες που να εξελίσσονται στη φάση αυτή και θα συγκεντρώσω την προσοχή μου στον ευρωπαϊκό μου προσανατολισμό και την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Τρεις φάσεις θα σημειώσω. Η πρώτη, μέχρι το 1990 μέχρι δηλαδή την πτώση του κομμουνισμού. Η δούλευα στο Υπουργείο ε, οικονομικού, ε, Εξωτερικού Οικονομικού Εμπορίου, ήμουν υπεύθυνο για τις σχέσεις ε, με τη Γερμανία και γενικότερα ασχολήθηκα με θέματα διεθνών σχέσεων και ασχολήθηκα γενικά με τις σχέσεις της χώρας μου με την Δύση. Έχω εξαιρετικές αναμνήσεις από όλες τις κοινέ προσπάθειες και τις επενδυτικές προσπάθειες τις οποίες συνεισέφερα και οι προσπάθειες αυτές εξακολουθούν να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Από το 1990 και μετά προσπάθησα να βοηθήσω την Ουγγαρία να ακολουθήσει το δρόμο που οδηγεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ η ατλαντική ολοκλήρωση και η ευρωατλαντική θα έλεγα ολοκλήρωση και πορεία της χώρας μου ήταν βασικός μου στόχος και γι' αυτό είχα διοριστεί και υπουργό Διεθνούς Εμπορίου. Και νομίζω ότι γενικά ο απολογισμός μου ήταν θετικός και αυτό το Ουγγρικό Υπουργείο είχε συγκεκριμένες οικονομικές και πολιτικές απόψεις οι οποίες είναι συμβατές θα έλεγα με την πορεία της χώρας. Μετά έρχεται η παρουσία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. έπρεπε από τη μία να βοηθάμε ε, την Ευρώπη να πάει μπροστά σαν ευρωβουλευτές αλλά και βασισμένοι στις εμπειρίες τις οποίες είχαμε σωρεύσει στο παρελθόν έπρεπε να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε και τις ευρωπαϊκές αξίες στην ίδια μου τη χώρα. Με την δεύτερη αυτή αποστολή θα έλεγα ασχολούμαι ακόμα και σήμερα με τη δική σας βοήθεια προωθώ τις ευρωπαϊκές αξίες και μπορώ να συνεχίσω να το κάνω όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και σε όλες τις υπηρεσίες των κρατών μελών. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε τον χρόνο που είχατε στη διάθεσή μας. Κυρία Γιάλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Φασάκα που είχαμε την τιμή και την τύχη να τον έχουμε ως ε, πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου. Και νομίζω ότι η περίοδος αυτή ήταν ακριβώς μία από τις ε, περιόδους όπου πετύχαμε τις περισσότερες αλλαγές και την περισσότερη πρόοδο τόσο όσον αφορά τις σχέσεις του Κοινοβουλίου με την Επιτροπή, με, με τον κύριο Κάλλας ε, που ήταν ο αρμόδιος επίτροπος και ακριβώς θεσπίσαμε ε, ένα στενότατο διάλογο και καταφέραμε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε πολύ περισσότερο τα μέσα ελέγχου της Επιτροπής μας αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι με τα ε, χάρη, όλα αυτά έγιναν και χάρη ε, στην ικανότητα του κυρίου Φασάκα, για να έχουμε αυτόν τον τόσο στενό διάλογο και τη συνεργασία με το ελεκτικό συνέδριο. Συνέβαλε λοιπόν και ο κύριος ε, Φασάκας στο να έχουμε αυτή την καλύτερη ε, περίοδο των σχέσεων μας με το ελεκτικό συνέδριο. Υπήρξε λοιπόν αυτή η καλή χημεία μεταξύ μα και αυτό οφείλεται και στον κύριο Φασάκα. Θα ήθελα λοιπόν να τον ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο απάντησε στι ερωτήσει αυτέ ο τρόπος με τον οποίο απάντησε δείχνει το ενδιαφέρον του για την ευρωπαϊκή υπόθεση γενικότερα και η προηγούμενη πορεία, πορεία του, ε, αυτό δείχνουν ότι θέλει να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του και τις γνώσεις του για να βελτιωθεί ε, ε, η αρμοδιότητα ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου σε αυτή τη νέα φάση στην οποία επισέρχεται το ελεκτικό συνέδριο. Θα ήθελα λοιπόν να μας ξεκαθαρίσετε το εξής. Το αναφέρεται και ταυτόχρονα ότι ε, ως πρόεδρος της ε, Κοκομπού και ακριβώς αναφερόμενος στις νέες βάσεις ε, συνεργασίας με το ελεκτικό συνέδριο, θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε τώρα λίγο περισσότερα και να εμβαθύνετε στο εξής. Ποιες, πώς βλέπετε το μέλλον και την δική σας ως μέλος υποψήφιο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ινέσα Σέντερ για την ερώτηση αυτή και για τα καλά της ε, λόγια για το έργο μου ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του και ε, μέλος του Κοινοβουλίου. Πριν από πέντε χρόνια προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την διαδικασία απαλλαγής ε, μαζί με τους συναδέλφους ε, τον κύριο Μόλτερ, ε, Καζάκα και την κυρία Κρέσλε. Με τους συναδέλφους αυτούς είχαμε στόχο την στενή συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο και επειδή ξέραμε τα προβλήματα έπρεπε να συνεργαστούμε στη μεταρρύθμιση της διαδικασίας απαλλαγής για να μπορέσει το ελεγκτικό συνέδριο να παρακολουθεί την διάθεση των κοντολίων και να έχει άποψη κατά διαδικασία απαλλαγής. Τα καταφέραμε λοιπόν να αλλάξουμε αυτή την ε, διαδικασία και μπορούμε να θεωρήσουμε επιτυχημένη την αλλαγή υπό το φως αυτών των ε, μεταρρυθμίσεων ενθαρρύναμε την καθημερινή συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο για να έχουμε αυτή την θετική διαβεβαίωση, τη θετική δήλωση εξοπιστίας όπως λέγεται και ε, φροντίσαμε να εμπλακούν και τα εθνικά κοινοβούλια και τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια που έχουν πάρα πολύ μεγάλη γνώση στον τομέα. Θα ήθελα εδώ πέρα να αναφερθώ στις πρόσφατες ε, θετικές εξελίξεις όταν το Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο προσπάθησαν να παλέψουν μαζί για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί καλύτερα, να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να δοθεί νέα ορμή στην ευρωπαϊκή οικονομία και φαίνεται πως ε, αυτό ακριβώς ε, θα είναι αποφασιστικό για τη συνεργασία ελληνικτικού συνεδρίου και κοινοβουλίου. κυρία Γιάλα. Σας ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φασάκας. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι ε, πρόκειτο για ένα ποιοτικό άλμα όσον αφορά αυτή τη νέα δυναμική συνεργασία με το Ελεκτικό Συνέδριο. Και βεβαίω εσεί συμβάλλατε ιδιαίτερα προ την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα επίση και με βάση τι απαντήσει σα να αναφερθώ στο εξή. Ακριβώ λαμβάνοντα υπόψη τα μέσα ελέγχου στα διάφορα κράτη-μέλη, θα ήθελα να σα πω ότι Εσεί μιλήσατε ε, για το γεγονό ότι στην Ουγγαρία το σύστημα ελέγχου δεν είναι παρόμοιο με αυτό που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να μου το αναπτύξετε λίγο περισσότερο αυτό το θέμα. Εφόσον ε, στο, στο, στη νέα φάση όλε οι πτυχέ των νέων μέσων και ε, η σχέση και ο συντονισμό με τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια θα ενισχυθεί ιδιαίτερα και με τα Εθνικά Κοινοβούλια βεβαίω. Λοιπόν, σας, ε, θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω, μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα ε, όσον αφορά τι ομοιότητε αλλά και τις διαφορές με το σύστημα ελεκτικού συνεδρίου στην Ουγγαρία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ο βασικός μας στόχος είναι να προωθήσουμε την στενή συνεργασία με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια γιατί έχουμε ένα κοινό καθήκον, τον έλεγχο και την παρακολούθηση του κοινοτικού προπολογισμού. Είχαμε πολλές ε, συναντήσεις ε, με την ε, Επίτροπη Επαφής και φροντίζαμε πάντα οι ελεγκτικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο να είναι συμβατές ή εναρμονισμένες έτσι ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών σε κάποια κράτη-μέλη ειδικά εκεί όπου υπάρχει περιφερειακή αυτονομία και εδώ πέρα βεβαίως αναφέρομαι στη Γερμανία εξεπλάγει πως ε, το Ομοσπονδιακό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπορούσε να πει στα ελεγκτικά συνέδρια, στα λέντερ, το τι ακριβώς θα κάνουν. Δεν υπήρχαν ενιαίες διαδικασίες. Αλλά είναι μια πρώτη προσπάθεια. Γι' αυτό ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να κάνουν εθνικές ε, δηλώσεις ε, για την χρήση του κονδυλίων και μετά διαπιστώσαμε πως σε κάποια κράτη-μέλη δεν ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο, αλλά βεβαίως το Ουγγρικό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Κόβατς ε, που με πρότεινε, άλλωστε, για αυτή τη θέση πρότεινε και κάποιες κοινέ μεθοδολογίες. Και όποτε η Ουγγρική κυβέρνηση, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στρέφονται σε αυτόν, με αίτημα ε, ελέγχου. Το Ουγγρικό Ελεγκτικό Συνέδριο απαντά ε, άμεσα παρά την ε, κάποια έλλειψη κονδυλίων. Ελπίζουμε λοιπόν γενικά να διαδοθεί αυτή η στάση και τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια να βοηθήσουν την διαδικασία απαλλαγής του Ευρωπαϊκού. Σας ευχαριστώ. Κύριος Ανδρέας, αν έχει το λόγο. Κυρία, συγγνώμη. Mr. Σας ευχαριστούμε κύριε Φασάκα που ήρθατε σήμερα. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτα απ' όλα, βλέπω στο βιογραφικό σας πως δεν έχετε εμπειρία. Καθόλου σχετική εμπειρία με τον έλεγχο. Στο παρελθόν η εμπειρία σας ε, είναι Πρόεδρο τη Επιτροπής Ελέγχου του προπολογισμού, αλλά από το εμπόριο και η μηχανία δεν έχει σχέση με αυτά. Οπότε πώς ε, θα αναλάβετε τέτοια ευθύνη όταν δεν έχετε τέτοια εμπειρία. Και το δεύτερο ερώτημα επίσης σχετίζεται με αυτό. Ήσταν πρόεδρος της Επιτροπής μας εδώ πέρα και τώρα θέλετε να γίνετε ελεγκτής. Το ερώτημά μου είναι εσείς θα δίνατε απαλλαγή στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για το 2008 με βάση την ε, γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας όταν λέτε ότι δεν έχω καμία εμπειρία σχετικά με τον έλεγχο το λογιστικό. Νομίζω ότι για πέντε χρόνια που ήμουν μέλος και πρόεδρος αυτής της Επιτροπής ασχολήθηκα με θέματα ελέγχου και επιθεωρήσεις λογιστικών. Ήδη από το 1981 πάντα ασχολήθηκα με τα οικονομικά. Πάντα ήμουν υπεύθυνο για να παρουσιάσω και να κάνω προτάσεις σχετικά με ελέγχους, ορκωτούς ή Ήμουν επίσης πολλές φορές μέλος ε, ελεγκτικών επιτροπών για διάφορες επιχειρήσεις που ανήκαν στα Υπουργεία στα οποία ήμουν υπουργό. Νομίζω ότι έχω εμπειρία που μου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσω να γίνω μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχει ξεκαθαριστεί άλλωστε ότι είναι προς όφελος ε, του ελεγκτικού συνεδρίου να έχει εκπροσώπους από όλες τις ε, επαγγελματικές δραστηριότητες, οικονομικούς εμπειρογνώμονες, γιατί ε, ακριβώς η διαδικασία ελέγχου γίνεται από επαγγελματίες ορκωτούς ε, ελεγκτές. Το προσωπικό δηλαδή είναι ορκωτοί λογιστές και νομίζω ότι οι επίτροποι είναι σε θέση να επιβλέψουν με την εμπειρία που έχουν αυτές τις δραστηριότητες. Έχω λοιπόν νομίζω την απαιτούμενη εμπειρία. Σχετικά με την απαλλαγή, μπορούμε να δώσουμε την απαλλαγή μόνο εφόσον υπάρχει θετική δήλωση. Μαζί με το ΣΥΜΚΑΛΑΣ ε, συνεργαστήκαμε ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κατεύθυνση αυτή. Εδώ και πέντε χρόνια Ε, τα αρνητικά σημεία ήταν πολλαπλάσια αυτών τα οποία συναντάμε σήμερα. Το 60% ήταν αμφισβητήσιμο σε επίπεδο εγκυρότητα στοιχείων, ενώ σήμερα αυτό το ποσοστό έχει κατέβει κάτω από το 30%. Βέβαια η απαλλαγή θα δοθεί δεν θα δοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορώ να δώσω εγώ απάντηση στο ερώτημά σας. Αυτό που βλέπω είναι ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν υπάρξει σημαντικές βελτιώσεις και είναι ρόλος και προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχίσει προς την κατεύθυνση αυτή. Η πρωτοβουλία της Ingeborg Γκρέσλε ήταν εξαιρετική στο παρελθόν. Ε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και για την εισαγωγή εσωτερικών ορκωτών ελέγχων και γενικά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα έλεγα είναι ανάλογοι των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και τα αποτελέσματα της προσπάθειας που κάνουν τα ευρωπαϊκά όργανα είναι ε, θετικά. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση λοιπόν αν θα δώσω ή δεν θα δώσω εγώ την ε, συγκεκριμένη απαλλαγή. Κύριος Χατζημαρκάκης, ευχαριστώ. Σε αντίθεση από την κυρία Αντρέασεν, εγώ θα ήθελα να πω πως χαίρομαι για το ότι θα ανήκει στο συνέδριο και κάποιος ο οποίος έχει πολιτική αντίληψη. Γιατί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται μόνο με τα νούμερα υπάρχουν, αλλά κάποιος πρέπει να κάνει και την πολιτική κρίση. Γι' αυτό χαίρομαι, κύριε Φαζάκας, που προταθήκατε εσείς. Ε, ενοχλήθηκα λίγο για αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος πριν από μισή ώρα γιατί πρέπει να πω πως ο κύριος Φαζάκας ε, είναι εδώ καιρό υποψήφιος, θα μπορούσαμε να ασχοληθεί πολύ νωρίτερα με την υποψηφιότητά του. Δεν είναι καλή αυτή η κίνηση και λυπούμε, ε, ε σέβομαι συνάδελφο, αλλά τώρα δεν είναι λογικό αυτό μισή ώρα εκ των προτέρων. Γνωρίζουμε ειδικά από τη Γερμανία τη δουλειά σας κύριε Φαζάκας, γι' αυτό μπορώ να πω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ικανότητά σας. Εγώ έχω μια πολύ απλή ερώτηση και γνωρίζω πως μπορείτε εύκολα να την απαντήσετε, αλλά απαντά, ε, αφορά με συγχωρείτε για τους υπόλοιπους συνυποψηφίους σας. Το θέμα των ξένων γλωσσών που υποτιμάτε, γιατί συχνά υπάρχει στο συνέδριο, υπάρχουν τρεις γλώσσες εργασίας και αν δεν τις ξέρει κανείς έχει πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Οπότε, πώς είναι τα αγγλικά και τα γερμανικά σας ή τα γαλλικά σας. Αυτή είναι η ερώτηση. Απαντά στα γερμανικά ο κύριος Φάζακας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν ναι, μου επιτρέπετε, είναι η πρώτη φορά που μίλησα Ούγγρικα. Ως πρόεδρος βεβαίως διήθυνα τις συνεδριάσεις Αγγλιστή Φάζακα. ήταν δυνατόν προσπαθούσα να μιλήσω γερμανικά. Και πραγματικά μου δίνει ουγγρικα ως πρόεδρο βεβαίω διηθυνα τη χαρά αυτό. Σήμερα το πρωί είχαμε και μια πολύ καλή ε, συνάντηση και τέθηκε αυτό το ερώτημα, μου είπαν τι γίνεται με τις τρεις ε, γλώσσες και πληροφορήθηκα με έκπληξη πως υπάρχουν μόνο τρεις, ε, τρεις δύο με συγχωρείτε, επίσημες γλώσσες ε, στο ελεγκτικό συνέδριο. Έτσι μου είπαν. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ πως είναι και οι τρεις γλώσσες εργασίας. όπως ξέρετε ήμουν πρέσβης ούτως ή άλλως Ουγγαρία στη Γερμανία. Θεωρούμουν ο κύριος Γερμανία στην Ουγγαρία. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, βεβαίω έχω σπουδάσει και αγγλικά. Εντάξει, εντωμεταξύ έχουν βεβαίω μειωθεί, αλλά νομίζω πως ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούγονται αγγλικά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαίω στα αγγλικά δεν είμαι στο ίδιο ακριβώς υψηλό επίπεδο με τα γερμανικά, αλλά είναι μια χαρά. Εντάξει, τώρα για τα γαλλικά δεν θα επιμείνω βεβαίω ότι έχω στο, το ίδιο επίπεδο, αλλά εν πάση Λοιπόν, για τις παρατηρήσεις σας, για την πολιτική αντίληψη. Προσπάθησα πολύ διπλωματικά να πω πως δεν ήμουν πολιτικός. Ήμουν πάντα τεχνοκράτης. Δεν ήμουν ε, μέλος του κόμματος πριν εκλεγώ ευρωβουλευτής και εντωμεταξύ βεβαίως δεν είμαι πλέον πια Μέλο του κόμματο. οπότε δεν έχω να παραιτηθώ από καμία θέση στο κόμμα, γιατί δεν είχα ποτέ τέτοια θέση στο κόμμα. Ήμουν σε διάφορα κινήματα υπέρ τη Ευρώπης, η Ουγγαρία στην Ευρώπη κτλ. Όλα αυτά ευρωκεντρικά. Νομίζω λοιπόν πως μιλάτε για αυτή την ε, πολιτική έποψη Κοιτάξτε, αν μιλήσουμε ότι έχω μια πολιτική άποψη, αυτό μπορεί να το κρίνω αρνητικά στην ε, Ουγγαρία. Εγώ θα έλεγα πως είμαι περισσότερο τεχνοκράτης. Τώρα, για αυτή την ε, κατηγορία εδώ πέρα, θα ήθελα να μου δώσετε λίγο χρόνο να σας πω πόσο τα πράγματα είναι εντελώς αντίθετα και ποιος ήταν ο πράκτορας. Ήμουν υπάλληλο του Υπουργείου που βεβαίως συνεργάζονταν με το Υπουργείο Ιστορικών. Όταν ετέθη το ζήτημα το 2002 λόγω του τότε Υπουργού μου ζήτησαν φακέλους, μου έδωσαν φακέλους από το Υπουργείο. Δείτε λοιπόν τα έγγραφα τα οποία τα έχουν ετοιμάσει άλλοι συνάδελφοι. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω καν τα ονόματά τους, αλλά αφορούσαν εμένα. Εγώ ήμουν το θύμα της παρακολούθησης και ζήτησα τότε επισήμως να δημοσιευτούν τα έγγραφα που με αφορούν για να δουν όλοι ότι πρόκειται περί διαπραγματεύσεων, περί τέτοιων θεμάτων, αλλά εγώ δεν... Ε, ε δεν μου έκαναν αυτή τη χάρη λόγω απορρίτου κτλ. Και, και ακόμα δεν έχουν δημοσιευτεί τα έγγραφα. Ο δε άνθρωπος ο οποίος με κατηγόρησε εμένα και τέσσερις άλλους βέβαια πρώην υπουργού ως ε, κατασκόπους ζήτησε εντωμεταξύ συγγνώμη βεβαίως. Τώρα για την άλλη υπόθεση ήμουν εκπρόσωπο, αντιπρόσωπος της Daimler Chrysler και είχαμε αγοράσει κάτι μηχανήματα από τη Ρωσία και ήταν ξεκάθαρο νομίζω πως η αγορά έγινε από την Ρωσία χωρίς να έχουμε εμείς κάποια εμπλοκή. Αμέσως το ίδιο απόγευμα ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος της Επιτροπής για την εμπλοκή του ονόματός μου. Και δεν νομίζω να έχουν σταθεί ποτέ αυτά σε κανένα δικαστήριο. Και κάτι ακόμα για το Υπουργείο μου. Το Υπουργείο μου θεωρήθηκε νομίζω θετικό τελικά και νομίζω πως ο κύριος Κόβατς κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια για να με προτείνει, για να πει πως πραγματικά και η εργασία του Υπουργείου μας ήταν υποδειγματική. Και είναι κρίμα που δεν είχα την δυνατότητα να απαντήσω νωρίτερα σε αυτές τις κατηγορίες, αλλά είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ kedves képviselőtársaim! Αγαπητά μέλη, από το 1988, πριν από την πτώση του κομμουνισμού, όταν ξεκίνησα την πολιτική μου δραστηριότητα, πάντα προσπάθησα να εκφράζω τις απόψεις μου υπέρ της Ενωμένης Ευρώπης. θεσμικά όργανα σαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν να παίξουν ένα, καλούνται να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και σήμερα στην επιλογή, στη διαδικασία επιλογής των, ε, των μελών του ελεγκτικού συνεδρίου. Το κοινό οφείλει να γνωρίζει το περιεχόμενο των συζητήσεων τις οποίες διεξάγουμε με τα υποψήφια μέλη μόνο μέσω ενός τέτοιου διαλόγου, μέσω ανοιχτού διαλόγου, μέσω της απόλυτης διαφάνειας μπορούμε να πάρουμε ενημερωμένες αποφάσεις. Πρέπει οι υποψήφοι να πληρούν τρεις προϋποθέσεις. Την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα και την ακαιρεότητα. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα σχετικά με την ακαιρεότητα σχετικά με τον κύριο Φαζάκας και γι' αυτό δεν τον θεωρώ κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση. Κοιτάξτε, εδώ δεν κάνουμε προσωπικές κριτικές. Είχατε δικαίωμα, όχι να κάνετε εκτιμήσεις, είχατε δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις. Η αξιολόγηση ακολουθεί. Εσείς ή θα θέσετε μία ερώτηση στον κύριο Φαζάκας ή όχι. Αν είναι κατάλληλος ή δεν είναι κατάλληλος ο κύριος Φαζάκας, αυτό θα το αποφασίσουμε σε ιστερότερη φάση. Περιμένω την ερώτηση. Τρεις ερωτήσεις θέλω να θέσω στον κύριο Φαζάκας. Η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών, της οποίας ήταν πρόεδρος, είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκε. Γιατί δεν είπε ότι από το 1976 μέχρι το 1989 ή το πράκτορ της μυστικής αστυνομίας της κομμουνιστικής Ουγγαρίας. Πρέπει να το παραδεχθεί ο κύριος Φαζάκας αυτό. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν μας ενημέρωσε ο κύριος Φαζάκας όταν έθεσε την υποψηφιότητά του για το ελεγκτικό συνέδριο ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια στην Ουγγαρία είχε εμπλακεί σε μία περίπτωση ε, διαφθοράς σχετικά με διεθνές εμπόριο όπλων. Και τρίτον, γιατί αρνείται ο κύριος Φαζάκας όταν ήταν υπουργό και υφυπουργό της Ουγγρικής κυβέρνησης, ότι κατά τη διάρκεια της υπουργίας του, το Ουγγρικό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν βρήκε κανένα πρόβλημα με τα οικονομικά του δικού του Υπουργείου, ενώ είναι δεδομένες οι πληροφορίες οι οποίες δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Υπουργείο αυτό υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα δυσδιαχείρισης. Λοιπόν, γιατί αρνείτε το ότι έχει υπάρξει μυστικός πράκτορ και γιατί αρνείτε το ότι έχει εμπλακεί σε μια περίπτωση διαφθοράς. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Φαζάκας, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να είναι σύντομοι. Αν ένας συνάδελφος μιλάει 4-5 λεπτά, οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις. Η ομιλία σας ήταν η τελευταία. Οι υπόλοιποι συναδελφοί σας δεν έχουν το χρόνο να θέσουν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όσον αφορά αυτές τις ερωτήσεις και οι τρεις ερωτήσεις στηρίζονται σε ισχυρισμούς τους οποίους απορρίπτω κατηγορηματικά και διαψεύδω. Δεν ε, υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ακαιρεότητά μου. Εγώ αυτό πιστεύω. Κοιτάξτε, ε, είναι, είναι κρίμα ότι αυτές τις πληροφορίες τις άκουσα πριν από μισή, ε, πριν από μισή ώρα. Όταν είχα, όταν είχα αναλάβει τα καθήκοντά μου, με, με, ε, ε, ε, υπέστην εξονυχιστικό έλεγχο όσον αφορά τα θέματα ε, εθνική ασφάλεια. Και μόλι θα γυρίσω στο σπίτι, θα στείλω στον κύριο Ντόιτ την έκθεση αυτή που αναφέρει ότι ποτέ δεν είχα αναμειχθεί με οποιοδήποτε τρόπο σε, σε υποθέσεις της μυστικής υπηρεσίας. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Συντερικών είχε φάκελο για μένα Κοιτάξτε, ε, πριν από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτο, αυτό ήταν σύνηθε για κάποιον υπουργό. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ήμουν πράκτορα μυστική υπηρεσία. Όσον αφορά την Daimler Κράισλερ, να σα πω το εξή. Εγώ επειδή η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας ασχολήθηκε με θέματα διαφθοράς, ε, εξέτασε την υπόθεσή μου, αλλά όταν ξεκαθάρισε την έρευνα μου ζήτησαν συγγνώμη και με απάλλαξαν από κάθε κατηγορία. Τρίτον, το Εθνικό Ελεκτικό Συνέδριο πάντα ε, μιλούσε με ιδιαίτερα θερμά λόγια και αναφερόταν με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη φοιτεία μου στο Υπουργείο. Αυτοί οι ισχυρισμοί ακούστηκαν το 2002. Ήμουν μέλος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνέχεια και πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν ξανάκουσα αυτές τις ε, ε υποτιθέμενες ε, περιπτώσεις ε, κακοδιαχείρισης από το 2002 και μετά ποτέ δεν άκουσα τίποτα. Εξάλλου, διακόπτω εντάξει, υπήρξε πρόβλημα με το μικρόφωνο. Ε, Κοίταξε, ακόμα και η αντιπολίτευση ε, με υποστήριξε και δέχτηκα τον ύψιστο έπαινο στη χώρα μου για την εργασία μου. Άρα λοιπόν δεν μπορώ παρά να επιβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ακαιρεότητά μου και πάντα βεβαίω να απαντήσω οποιαδήποτε περαιτέρω ερώτηση. Τελευταία ερώτηση για 30 δευτερόλεπτα, γιατί πραγματικά είμαστε εκτό χρόνου. Κρέσλε Ευχαριστώ και καλώ ήρθατε κύριε Φαζάκα. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και καλό είναι επιτέλους να τελειώσει αυτή η υπόθεση με αυτές τις κατηγορίες γιατί πρέπει να συνεργαστούμε στο μέλλον. Οπότε το ερώτημα μου είναι τι μπορούμε να, περιμένουμε από σας. Αλλιώς νομίζω πως γνωριζόμαστε ήδη αρκετά καλά και είστε ένας από τους λίγους που ξέρει τα πράγματα και από τη σκοπιά του Κοινοβουλίου. Και καλό θα ήταν πια να ξεκαθαρίσουν αυτές οι κατηγορίες. Να θέσω εγώ ένα ερώτημα. Οπωσδήποτε θα κάνω μια δήλωση. Ναι, ναι. Ευχαρίστως θα αντικρούσω αυτές τις κατηγορίες. Ίσως σήμερα κιόλας. Αλλά νομίζω πως πρέπει να γραφτούν στα πρακτικά αυτά τα οποία είπα για αυτές τις κατηγορίες. Ακόμη λοιπόν μια φορά κυρία Γκρέσλε, γνωριζόμαστε καιρό και ποτέ δεν είχε αναφερθεί πως το 2002 υπήρχε αυτό το περιστατικό και με πολλές άλλες ε, υψηλές ε, προσωπικότητες ε, οι οποίες χειρίζονταν φακέλους στο... και είχαν φακέλους, κρατούσαν φακέλους για αυτούς στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν σημαίνει πως κάποιος ο οποίος δουλεύονταν σε μια, σε μια πρεσβεία δεν καταγράφονταν οι δραστηριότητες του. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασά Φαζάκας για την ακρόαση και περνάμε στην επόμενη ακρόαση του επόμενου υποψηφίου για το ελεκτικό συνέδριο από τις τηλεφωνικές αρχές, την κυρία Ράσα Μπουτμπεργκίτε. úr, csak a későbbi véget, Πρόεδρε, για να αποφύγουμε ε, κάποια παρεξήγηση, εάν μπορούμε να αποδείξουμε ότι ο κύριος Φαζάκας δεν είπε την αλήθεια, εάν αν αποδείξω ότι ε, ε ψεύδεται, τι θα γίνει, θα επανέλθουμε αύριο μπορούμε να έχουμε κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ. Το είπα και προηγουμένω. Όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, θα τα συζητήσουμε αύριο, όταν θα περάσουμε στη φάση τη αξιολόγηση. Ε, σήμερα ε, έχουμε μόνο τι ακροάσει. Ερωτήσει, απαντήσει και παρουσίαση του ηγητή. Σα παρακαλώ, έχετε το λόγο. Eh, Καλώς ορίσατε λοιπόν. Να σας πω ότι έχετε πέντε λεπτά. Καλησπέρα σας λοιπόν. Πέντε λεπτά για την αρχική παρουσίαση. Στη συνέχεια θα έχουμε δέκα λεπτά ερωτήσεις από την εισηγήτρια και στη συνέχεια ε, τις ερωτήσεις των υπολείπων ε, μελών της Επιτροπής. Έχετε το λόγο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 Κυρίες ε, και κύριοι, είναι τιμή μου και ευχαρίστηση να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας και να συζητήσουμε πώς θα συνεισφέρω σε πιο σε, έναν πιο αποτελεσματικό, σε μια πιο αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης εάν γίνω μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το 2006 είχα ήδη το προνόμιο να βρεθώ ενώπιον της Επιτροπής έλεγχου του προϋπολογισμού να μοιραστώ τις εμπειρίες μεταξύ του Λιθουανικού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα της Επιτροπής Μουσιονομικού Ελέγχου και του δικού μας ελεγκτικού συνεδρίου για το πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε ορθά τα δημόσια οικονομικά. Και είμαι λοιπόν πεπισμένη πως η σημερινή ακρόαση είναι μια καλή ευκαιρία για να έχουμε μια μακρόχρονη συνεργασία. Όλη μου η σταδιοδρομία ήταν στο δημόσιο τομέα, ήμουν διοικητικός παλαιός σε πολλά Υπουργεία και στο Ελληνικό Συνέδριο και ασχολούν με θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση δημοσίων οικονομικών και τον έλεγχο. Και αναμένω λοιπόν πως η επαγγελματική μου επάρκεια είναι επαρκής και η εμπειρία μου επίσης θα μου επιτρέψει να αναλάβω τα καθήκοντα του μέλους του Ελληνικού Συνεδρίου όπως τα ορίζουν οι συνθήκες. Πιστεύω πως οι αξίες ε, τις οποίες ακολούθησα για πολλά χρόνια μου δίνουν ε, την δυνατότητα να αντιληφθώ τις προσδοκίες των ανθρώπων για το πώς θα λειτουργήσει καλύτερα το ελεγκτικό συνέδριο. Ήμουν πάντα ανεξάρτητη και αμερόληπτη. Θα ήθελα λοιπόν να σας διαβεβαιώσω πως στην περίπτωση στην οποία οριστώ μέλος του ελεκτικού συνεδρίου θα βασιστώ στην ανεξαρτησία και στα λογιστικά, τα ελεγκτικά πρότυπα και θα ακολουθήσω βεβαίω τις ε, απαιτούμενες προδιαγραφές. Θα κινηθώ σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα θα ακολουθήσουμε αυστηρά τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και πρακτικών που έχει ορίσει το συνέδριο. Δεύτερον, θα εργαστώ αποτελεσματικά σε όλες τις ιδιότητες που θα έχω και θα φροντίσω να δρω προληπτικά έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους στρατηγικούς στόχους του συνεδρίου δηλαδή να έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα οι έλεγχοι και να είναι πιο αποτελεσματικοί Κατά την άποψή μου, το συνέδριο θα πρέπει να υποστεί τις εξής βελτιώσεις, να υπάρξει έλεγχος ποιότητας και διασφάλιση ποιότητας, καλύτερη χρήση των πόρων και να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι της λειτουργίας. Είμαι εγώ υπέρ της ανοιχτής συνεργασίας. Θεωρώ πως το συνέδριο θα πρέπει να βελτιώσει τη συνεργασία με την Κομισιόν και τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Στην δε πρώτη περίπτωση χρειαζόμαστε συνεργασία με την Κομισιόν για να μην γίνονται δύο φορές τα ίδια πράγματα και να μην υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες και επίσης η συνεργασία μεταξύ του συνεδρίου και του κοινοβουλίου είναι ουσιαστική και αυτό το ξέρω γιατί είχα δουλέψει πέντε χρόνια στο κοινοβούλιο μόνο εάν υπάρχει ένας κύκλος λογοδοσίας όπου όλοι ξέρουν τις ευθύνες τους ε, και δρούν αποφασιστικά θα θέσει τους όρους για καλύτερη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Υποστηρίζω πλήρως λοιπόν τις προτάσεις σας για να οργανωθεί μια συζήτηση για τις εθνικές δηλώσεις, ε, τις διαβεβαίωσεις αυτές τον ε, κίνδυνο του ανεκτού σφάλματος ε, και την απλοποίηση των κανόνων. Τα ερωτήματα αυτά εκκρεμούν εδώ και καιρό στις ε, συνεδριάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου και όμως δεν έχουν ακόμα απαντηθεί. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ε, είμαι ικανοποιημένη που έχω αυτή την ευκαιρία για να σα διαβεβαιώσω πως εγώ θα ήθελα να μπορέσουμε να ζητήσουμε από κοινού απαντήσεις. Θα σας ακούσω προσεκτικά καθώς εκπροσωπείτε τους πολίτες της ΕΕ, Ευρώπης, ε, τις ανάγκες τους και τις φιλοδοξίες τους και ελπίζω έτσι να συνεισφέρω στο έργο του ελεγκτικού συνεδρίου που είμαι πεπισμένη είναι ένα από τα όργανα ελέγχου με το μεγαλύτερο επαγγελματισμό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω τις ερωτήσεις σας. Η συγγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Είσαστε νομίζω ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο από υφυπουργό μπορούμε να γίνουμε μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Οι απαντήσεις τις οποίες θα μας δώσετε, ήταν, τις οποίες μας δώσατε μάλλον που ακούσαμε, ήταν ικανοποιητικές. Εσεί αναφερθήκατε σε απαντήσει στο γεγονό ότι το 80% του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αντικείμενο διαχείριση μέσω τη ε, κοινή τη ε, διαχείριση. Και υπάρχει μια έλλειψη συνημετρία βεβαίω, διότι η ευθύνη για τον έλεγχο ανάμεσα στο ελεκτικό συνέδριο ε, και τα εθνικά όργανα ελέγχου δεν υπάρχει ακόμα, αν θέλετε. Λοιπόν, σε ρωτώ, τι σκέφτεστε να κάνετε κατά τη διάρκεια της ε, θητείας σας, αν έχετε κάποια ιδέα. Επίσης βλέπω ότι ε, αναφέρεστε στο γεγονό ότι από την 1η ε, ε, Ιανουαρίου στο 2010 ε, ότι το γραφείο σας ε, ε, κάνει follow-up των ελέγχων. Μα και εμείς θέλουμε να συμπεριλάβουμε αυτή την ιδέα και να γίνεται όλο και περισσότερο από το ελεκτικό συνέδριο. Σας ρωτώ λοιπόν, μήπως έχετε κάποια ιδέα που θα μπορούσατε να προτείνετε όσον αφορά τη δάση των αρμοδιοτήτων σας ως υποψήφιο μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι η ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ε, μοιράζεται ανάμεσα ε, ε, στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη, αλλά η ευθύνη δεν μοιράζεται εξίσου. Ε, και υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται και από τη συνθήκη. Σήμερα δεν μπορώ να πω ότι τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να ε, δεν μπορούν να αλλάξουν τις ε, διατάξεις της συνθήκης. Ε, δεν έχουν αυτήν την αρμοδιότητα. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης των δραστηριοτήτων ελέγχου και των δράσεων ελέγχου που λαμβάνουν χώρα στα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και εδώ αναφέρομαι στη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και στην επαλήθευση των διαφόρων οικονομικών συναλλαγών. Ε, καθώς επίσης και στο, στον έλεγχο του κατά πόσον τα ε, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά. Τα ε, το ελεκτικό συνέδριο θα μπορούσε να συνεργαστεί με, τους, με, με τα αρμόδια όργανα ελέγχου των κρατών μελών. Βεβαίω γνωρίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, να μην πω αδύνατο, το ελεκτικό συνέδριο να αναλάβει ε, τη δράση του βασικού ελέγχου. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο, ε, δεν είναι εύκολο πάντα να παρακολουθηθούν τα αποτελέσματα των εθνικών ελέγχων. Αλλά εδώ έχουμε τις ε, διατάξεις της συνθήκης. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να σκεφτούμε το πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τα κονδύλια αυτά και, εγώ θέλω να συμβάλλω, και του πόρους που έχουμε στη διάθεσή μα. Εγώ θέλω να συμβάλλω προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, κυρία Γιάλα, Σας βλέπω ε, γεμάτη ε, καλών προθέσεων, αλλά τα πράγματα είναι όλο και περίπλοκα κάθε μέρα. Λοιπόν, εσεί στο ερωτηματολόγιο και στην απάντησή σας αναφέρεστε στην ανάγκη υπέρβασης αυτού που μέχρι στιγμής υπήρξε καθαρά τεχνοκρατική προσέγγιση. Και πιστεύετε, τουλάχιστον αυτό φαίνεται μέσα από τι απαντήσει σας, ε, πιστεύετε ότι πρέπει να προωθηθεί η ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, ανάλογα φυσικά με τι αρμοδιότητε του καθένα και με το ρόλο του για να έχουμε ένα σύνολο ε, διαχειριστικής ε, νοοτροπίας αν θέλετε. Όλα αυτά όμως τι είναι, είναι καλές προθέσεις ή υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχετε ξεκάθαρες ιδέες για το πώς από αυτή την προσέγγιση την καθαρά τεχνοκρατική την οποία εσείς επικρίνετε θα μπορούσαμε να περάσουμε μέσα σε μια ε, πραγματικότητα ενθουσιώδους συμμετοχής, γιατί σε αυτό το επίθετο χρησιμοποιείτε όλων των εμπλεκομένων για ένα απολύτως αυστηρό αλλά και αποτελεσματικό έλεγχο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά ότι η συνθήκη της Λισαβόνας προτρέπει ιδιαίτερα τη συνεργασία ανάμεσα στο ελεκτικό συνέδριο και τα εθνικά όργανα. Αλλά η ευθύνη του ελέγχου ανήκει στο ε, ελεκτικό συνέδριο. Πιστεύω, και τουλάχιστον αυτό μπορώ να πω με βάση τη δική μου την εμπειρία, ότι δεν υπάρχει πάντα αμοιβαία κατανόηση του, της σημασίας της χρησιμοποίησης των πόρων με τον βέλτιστο τρόπο. Και όταν μιλώ εδώ ότι δεν υπάρχει αμοιβαία κατανόηση, αναφέρομαι στα εθνικά όργανα ελέγχου και στο λεπτικό συνέδριο. Ο στόχος μας ποιος είναι, να, να κατανοήσουμε όλοι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου μπορούν να αξιοποιηθούν. Και ο βασικός ελεγκτής, εμπροκειμένο το Ελεκτικό συνέδριο, θα μπορούσε να αξιοποιήσει την εργασία των εθνικών οργάνων ελέγχου, αλλά ε, παρέχοντας την απόδειξη ότι ο έλεγχος στηρίζεται σε έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία. Στο Ελεκτικό Συνέδριο, μια ομάδα εργασία ε, μελετά ε, το θέμα αυτό και κινείται προς την κατεύθυνση που σας ανέφερα και εγώ. Ο στόχος είναι η εισαγωγή κάποιων αλλαγών στην ε, δομή ε, των ε, δηλώσεων εξακρίβωσης έτσι ώστε να υπάρξει, ε, να υπάρξει ένα σωστό σύστημα. Ε, και ε, όσον αφορά αυτές τις δηλώσεις αξιοπιστίας, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. και τα αποτελέσματα και θα πρέπει να εξεταστούν τα ευρήματα του ελεκτικού συνεδρίου. Πάντως σήμερα δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να σας πω πιο συγκεκριμένα τι θα έκανα εγώ αν ήμουν μέλος του, του ελεκτικού συνεδρίου. Αυτό που πιστεύω πάντως είναι ότι θα πρέπει από κοινού να ψάξουμε να βρούμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. θα πρέπει να έχουμε σαφή εργαλεία έτσι ώστε να είμαστε ε, περισσότερο νόμιμοι αλλά και αποτελεσματικοί όσον αφορά την χρήση των ε, κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, θα παρακαλούσα την ε, ομιλήτρια να είναι πιο συνοπτική στι απαντήσει γιατί έχουμε πολλέ ερωτήσει. Κυρία Γιάλα, 30 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, εσεί μιλήσατε για τη συνεργασία και την ανταλλαγή ε, απόψεων σε, σε συνεχιζόμενο επίπεδο και στοιχείων ανάμεσα στα εθνικά ελεκτικά συνέδρια και στο ελεκτικό συνέδριο. Εγώ όμω θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Τι γίνεται με την ανεξαρτησία όλων των οργάνων και των μεν και των δε. Απάντηση. Κοιτάξτε, η συνθήκη, η συνθήκη προβλέπει υποχρέωση συνεργασίας μεταξύ του ελεκτικού συνεδρίου και των εθνικών ελεκτικών οργάνων και ταυτόχρονα διασφάλιση της ανεξαρτησίας όλων. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι γνωρίζω με βάση την εμπειρία μου τι σημαίνει η λέξη ανεξαρτησία. Και να σας πω και το εξής, ίσως σήμερα δεν είναι όσο στενή θα έπρεπε η συνεργασία, επειδή ακριβώς το κάθε όργανο ε, έχει ακριβώς στο μυαλό του την έννοια της ανεξαρτησίας και δρά ε, με σκοπό τη διασφάλιση της αρχής αυτής. Τώρα όμως θα πρέπει να είναι πιο ε, ε, καρποφόρα η συνεργασία ανάμεσα στο Ελληνικό συνέδριο και στα φοινικά όργανα. Πιστεύω ότι η λέξη ανεξαρτησία είναι η πιο σημαντική αρχή που θα πρέπει να διασφαλίζεται από κάθε ανώτατο όργανο ελέγχου. Βεβαίω ε, δεν είναι μια απόλυτη αρχή, διότι κάθε όργανο, ενώ διασφαλίζει την ανεξαρτησία του, θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι υπόλογο σε κάποιον άλλον. Γιατί και η αρχή τη λογοδοσία είναι πολύ σημαντική. Πρώτα απ' όλα ενώπιον των πολιτών μα. ή στου ε, ερετού εκπροσώπου, όπω τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία μας και ταυτόχρονα πιστεύω ότι οι εθνικοί ελεκτές και το ελεκτικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πάνω απ' όλα τις προσδοκίες, κυρίως τις νόμιμες προσδοκίες των πολιτών. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι σε αυτή τη φάση δεν θα πρέπει να βιαστούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να εκφράσω μια άποψη η οποία είναι πολύ θετική για την υποψήφια, τη Βασαμπουμπεργίτε. Έχει πράγματι πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, όχι μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά πάντως τουλάχιστον αυτά τα πέντε χρόνια κατάφερε να δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό και καινοτόμο σύστημα ελέγχου στη χώρα. Με υψηλής ποιότητας ελέγχου, με καλό και επαρκές προσωπικό ε, και πλήρως αποπολιτικοποιημένη υπηρεσία και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και είναι επίσης και η μόνη γυναίκα ανάμεσα στους εννέα υποψηφίους για το ελεγκτικό συνέδριο. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ανησυχούμε για το πώς θα χρησιμοποιηθούν σωστά τα χρήματα του Ευρωπαίου πολίτη. Κατανοώ την ε, ερώτησή σας, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Θα ήθελα να μην αναφερθώ αναλυτικά στα θέματα της μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής πολιτικής ή της μεταρρύθμισης της κοινή αγροτικής πολιτικής και να μην μιλήσω και για την εφαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού. Θα ήθελα όμως να εκφράσω την άποψη του Ελεκτικού συνεδρίου του 2009 για την εφαρμογή του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιολόγηση που γίνεται για τον προϋπολογισμό αυτό είναι μια θετική αξιολόγηση επισημένονται όλες οι θετικές τάσεις οι οποίες είχαν υπογραμμιστεί στο παρελθόν σχετικά με τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Είναι σαφές επίσης ότι παραμένουν ορισμένα προβλήματα σε εκκρεμότητα τα οποία δεν είναι τόσο θετικά όσο εμείς θα επιθυμούσαμε ότι ήταν κάποιες από τις ενέργειες οι οποίες εγκρίνονται δεν είναι οι σωστές, δεν είναι επίσης νομότυπες. Όπως ίσως γνωρίζετε, θα πρέπει να αναφερθούμε πιο ειδικά στο Ταμείο Συνοχής. Μιλάμε για το 1 τρίτο περίπου του κοινοτικού προϋπολογισμού και αυτός είναι ένας χώρος στον οποίο σωρεύονται πάρα πολλά από τα προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, άνω του 10%. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό το 11% είναι ανυπόφορα υψηλό επίπεδο. Και γι' αυτό το ελεγκτικό συνέδριο κάνει σε αιτήσια, σε αιτήσια βάση ορισμένες συστάσεις για τη βελτίωση των ελεκτικών μεθόδων. Νομίζω ότι οι συστάσεις αυτές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο από τον ένα χρόνο στον άλλο και να εκφράσω εδώ την ευαρέσκειά μου ε, για τις προσπάθειες τις οποίες έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη για τη συνεχιζόμενη βελτίωση του συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δάσης, το οποίο όμως καλεί να υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες για βελτίωση. Οι κανόνες ε, με τους οποίους κινούμε θα είναι περίπλοκοι και είναι απαραίτητο να απλοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες ιδιαίτερα σχετικά με την επιλεξιμότητα ορισμένων προτινομένων για χρηματοδότηση προγραμμάτων. Επίσης ε, ε, ελείπουν ορισμένα κριτήρια τα οποία είναι σημαντικά. Πρέπει λοιπόν να απλοποιήσουμε τους κανόνες για να καταστήσουμε τα συστήματα ελέγχου κατανοητά σε όλους και να διασφαλίσουμε την νόμιμη χρήση ε, των κοινοτικών ποσών. Κύριε Σένα. Η προϋπηρεσία σας στο Γενικό Ελεγκτικό Συνέδριο της Λιθουανίας είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό και νομίζω ότι θα αποδώσετε πολλά σαν μέλος και πράγματι ελπίζω να συνεργαστούμε στο ΣΤΑ στενά στο μέλλον. Αναφερθήκατε στις ανεξάρτητες ε, εκτιμήσεις. Ποια είναι η άποψή σας για το ότι το ελεγκτικό συνέδριο είναι ένα επιπλέον κοινοτικό όργανο το οποίο χρηματοδοτείται από τον ίδιο προϋπολογισμό με τα άλλα όργανα. Μπορείτε να πιστέψετε ότι ένα τέτοιο όργανο είναι ανεξάρτητο. Σχετικά τώρα με τις εκφράσεις τις οποίες χρησιμοποιήσατε απαντώντας στην απάντηση 7 ότι δεν θα δεχθείτε καμία υποχώρηση στην νομοτυπία, παρατυπία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απατών και διαφθοράς. Πιστεύετε ότι η παρούσα ντάς, η δήλωση αξιοπιστίας δηλαδή είναι μια συμβιβαστική λύση σε επίπεδο αξιοπιστίας. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού ε, δεν έχει λάβει θετική κρίση και εσείς σαν ελέγκτρια νομίζω μπορείτε να κατανοήσετε που είναι το πρόβλημα. Η τρίτη ερώτηση. Θα κάνετε ό,τι προσπάθειες περνάνε από χέρι σας έτσι ώστε ε, να δημοσιοποιηθούν όλα τα οικονομικά συμφέροντα των μελών του ελεκτικού συνεδρίου όπως συμβαίνει με τους επιτρόπους. Η ερώτηση σχετική με την ανεξαρτησία του ελεγκτικού συνεδρίου της υπηρεσίας ε, επειδή ε, εξαρτάται από το εκτελεστικό αν θέλετε κομμάτι της εξουσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μου. Ε, το, το Γενικό Λογιστήριο το οποίο ασκεί ελεγκτικές δραστηριότητες χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση. Είμαστε λοιπόν εν μέρη εξαρτημένοι από το Υπουργό Οικονομικών, αλλά σύμφωνα με την εμπειρία που έχω μέχρι τώρα να σας διαβεβαιώσω ότι ε, το ελεγκτικό συνέδριο το ευρωπαϊκό χρηματοδοτείται και δεν επηρεάζεται από τα όργανα τα οποία συνεισφέρουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Σέβομαι ιδιαίτερα όλα τα παλιά κράτη-μέλη στα οποία τα ελεγκτικά συνέδρια ε, χρηματοδοτούνται άμεσα χωρίς να περνούν από τις υπηρεσίες της πολιτικής ε, κυβέρνησης, διακυβέρνησης γιατί αυτό διασφαλίζει περισσότερη ανεξαρτησία. Παρακολουθώ τις δηλώσεις αξιοπιστίας από το ελεγκτικό συνέδριο τον τελευταίο καιρό και βλέπω τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία καταθέτει σε αιτήσια βάση το ελεγκτικό συνέδριο και είμαι πεπισμένος ότι το συνέδριο αυτό είναι απολύτως ανεξάρτητο και σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από το δημοσιονομικό τρόπο χρηματοδότησής του. Να σας διαβεβαιώσω επίσης ότι κάθε μορφή διαφθοράς και κάθε μορφή απάτης που θα μπορούσε να υπάρξει είναι κάτι το οποίο θα απειλήσει τη δημοκρατία και την ανάπτυξη κάθε χώρας και κάθε συνόλου χωρών. Όπως σας είπα εργάζομαι στον δημόσιο τομέα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πάντα ήμουν κατά κάθε τάσης η οποία θα οδηγούσε σε απάτες και σε διαφθορά. Είμαι πεπισμένη ότι όταν υπάρχει διαφθορά σε εθνικό επίπεδο ή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν υπάρχουν παρατυπίες έστω, πρέπει να αντιμετωπιστούν αμέσως και γι' αυτό μειώνεται ο αριθμός τους με τον καιρό. Προφανώς και υπάρχουν πάντα προβλήματα και γι' αυτό εμείς καλούμεθα να ασκήσουμε τις αρμοδιότητές μας. Και υπάρχουν φυσικά και τα λογιστικά επίπεδα τα διεθνή συγγνώμη λογιστικά επίπεδα τα οποία θα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Θυμίζω ότι εμείς δεν έχουμε σαν στόχο την καταπολέμηση της, απάνης, της ε, απάτης. Συγγνώμη. Υπάρχουν υπηρεσίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά αυτό ουσιαστικά κάνει ο κάθε, το κάθε μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου έτσι ώστε να μην φύγονται τα συμφέροντα της δημοκρατίας και των πολιτών. Σχετικά με την τρίτη σας ερώτηση, φυσικά και είμαι διαθέσιμη να δηλώσω όλα τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία έχω εγώ και η οικογένειά μου και να σας διαβεβαιώσω ότι προς στιγμή. επειδή είμαι υπεύθυνη για το ελεγκτικό συνέδριο της Λιθουανίας, ε, τα οικονομικά μου δεδομένα και τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία έχω εγώ και η οικογένειά μου δημοσιοποιούνται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι και πάλι αφορά τις γνωσικές σας ε, γλώσσες. Κάντε μια δήλωση στα αγγλικά, καλό αυτό. Αν μπορείτε να απαντήσετε και στα αγγλικά ή στα γαλλικά, καλό θα ήταν. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, ο οποίο προβλέπεται στην ε, συνθήκη της ε, Λισαβόνα Υποστηρίζετε ένα τέτοιο μέσο και ω ελεγκτικό συνέδριο θα συνεργαζόσασταν με τον ε, Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ευχαριστώ. Yes. Ναι, πράγματι, προβλέπει αυτή την δυνατότητα η συνθήκη περί ενός Ευρωπαίου εισαγγελέα ή μιας Ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Και εγώ είμαι υπέρ οποιασδήποτε ιδέας σημαίνει περισσότερη λογοδοσία για να βρούμε τις ε, και να αντιμετωπίσουμε τις παρατυπίες. Αλλά φοβάμαι λίγο πως δεν θα είναι τόσο εύκολο να βρούμε κοινέ λύσεις για 27 κράτη-μέλη, γιατί είναι μόνο δυνατότητα η οποία δίνεται. Και ίσως θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερη βάση στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ Όλαφ, Eurojust και εθνικών ε, θεσμικών αρχών και κυρίως οργάνων επιβολής της τάξης. Ο, ο κύριος Ντόιτς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά εδώ δεν έχουμε χρόνο. Και μιλάμε ταυτόχρονα πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα. Πώς λοιπόν να θέσει κανείς σε 7 δευτερόλεπτα μια ερώτηση και να, η οποία θα πρέπει να απαντηθεί σε τέσσερα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, εντάξει, προσπαθώ να είμαι πολύ σύντομο. Δύο ερωτήσει έχω. Πρώτη ερώτηση. Ποιε είναι οι τομεί ε, του, ευρωπαϊκού, ε, του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζονται αυστηρότερο έλεγχο στα προσεχή χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, αναφέρατε ότι η νέα δημοσιονομική πολιτική ε, ξεπερνά τα πλαίσια της συγκεκριμένης ακρόασης. Όμως, η τεράστια πύρα του ελεκτικού συνεδρίου, κατά την άποψή σας, θα μπορούσε να τεθεί ε, στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια συζήτηση. και σε ποιο βαθμό, ε, και ανάλογα βέβαια και με το βαθμό που θα συμμετάσχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και το ε, Συμβούλιο προς την δημοσιονομική μεταρρύθμιση. Και βεβαίω χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε και μία γυναίκα υποψήφιο, κυρίω που είχαμε και την Παγκόσμια ημέρα γυναίκα 8 Μαρτίου. Όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα, θα ήθελα να σας παραπέμψω στην ε, ε, τελευταία ειδική έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου όπου εντοπίστηκαν οι βασικοί τομείς κινδύνου. Συμφωνώ με την ε, άποψη αυτή, με την άποψη του Ελληνικού Συνεδρίου, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα ελέγχου. Στη συνέχεια, όσον αφορά τον, το επίπεδο του ανεκτού κινδύνου, θα πρέπει να δούμε το κόστος του ελέγχου. Για, για παράδειγμα, όταν μιλάμε για ε, τη συνοχή ή τα, ή τα, γεωργικά ζητήματα. στην μία περίπτωση ε, το κόστος αυτό είναι 4%, στην άλλη 0, κάτι. Άρα λοιπόν πρέπει να ληφθούν όλα αυτά υπόψη. Και κάτι άλλο το οποίο ήδη ανέφερα και το οποίο θα ήθελα να παραλάβω, είναι το εξή. Θα ήταν σωστό να απλοποιηθούν οι κανόνες, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιλεξιμότητα. Και θα ήταν επίσης φρόνιμο να συνεργαστούμε ιδιαίτερα στενά με τα κράτη-μέλη, γιατί οι περισσότερες παρατυπίες προέρχονται από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Και εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να καταβληθούν οι περισσότερες προσπάθειες. Τώρα, όσον αφορά το πώς θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την πιο αποτελεσματική, ε, το πώς θα δαπανώνται τα χρήματα πιο αποτελεσματικό τρόπο και ότι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνται νόμιμα και αποτελεσματικά, να είμαστε σίγουροι ότι πρώτα απ' όλα ε, υπάρχει διάλογος και στη συνέχεια να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι ε, για κάθε καινούρια δημοσιονομική ε, περίοδο. Και όπως ανέφερε και στην τελευταία ειδική έκθεση το ελεκτικό συνέδριο, τώρα βρισκόμαστε το 2010 και ήδη θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ε, το επόμενο χρονικό διάστημα, από 2014 και εξή. Και εδώ ε, θα ήθελα να σας πω ότι με βάση την εθνική μου επαγγελματική εμπειρία, ε, το χρονικό διάστημα από 2007 στο 2013 δεν είχε, δεν είχε υποστεί τη σωστή προετοιμασία. Και όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα, δεν υπήρχε ο κατάλληλος βαθμός προετοιμασίας στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι μετά την ε, πρώτη είστε η δεύτερη γυναίκα από την Λιθουανία. Βέβαιως ε, κάθε μία είναι διαφορετική και όσον αφορά τη συνεργασία μας θα ήθελα να σας ρωτήσω η Λιθουανία είναι δύσκολη περίπτωση όσον αφορά την διαφθορά. Εάν δούμε το βαρόμετρο της διεθνούς διαφάνειας, η Λιθουανία είναι σε ηγετική θέση. Εσείς τι έχετε κάνει μέχρι στιγμή στα διοδρομία σας για να αντιμετωπίσετε ε, αυτό το, το θέμα, ποιο είναι το σημαντικότερο επίτευγμα το οποίο μπορείτε να μας αναφέρετε. Η υπηρεσία σχετική στη Λιθουανία δεν είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Έχουμε δύο φορείς ε, στην Λιθουανία, την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων που ασχολείται με τη διαφθορά και την Υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος που ασχολείται με την απάτη. Το δε ελεγκτικό συνέδριο έχει συμφωνίες ε, με αυτούς τους δύο φορείς και συνεργαζόμαστε. Η μεγαλύτερη επιτυχία που μπορώ να αναφέρω είναι η εξής όλα τα υλικά τα οποία μεταφέρονται από εμάς στην υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος ερευνώνται και πολύ συχνά ο Όλαφ παρακολουθεί αυτές τις ε, περιπτώσεις και πράγματι έχουμε διαπιστώσει κάποιες περιπτώσεις ε, απάτης. Είχαμε λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες ε, οι ελεγχόμενοι είχαν ε, χρησιμοποιήσει κονδυλία Σάπαρτ και είδαμε πως υπήρχε κάποια απάτη, δώσαμε τα υλικά στην υπηρεσία δίωξη οικονομικού εγκλήματος και πράγματι όλα επιβεβαίωσε ότι υπήρχε απάτη. Υπήρχε μια εταιρεία η οποία υπέβαλε πλαστά έγγραφα και αναγκάστηκε βεβαίω να ε, επιστρέψει τα κονδύλια αυτά. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει νομίζω και μια δικαστική απόφαση του μεταξύ Λιθουανία. Έχει ε, καταλήξει τίποτα στα δικαστήρια. Ε, ακούστε, έχουμε τα ίδια δικαστήρια, το ίδιο σύστημα ε, στη Λιθουανία όπως σε κάθε άλλη δημοκρατική χώρα έχουμε δικαστήρια ποινικά και διοικητικά. Και οι περιπτώσεις ε, διαφθοράς ε, και απάτης βεβαίως αφορούν τα ποινικά δικαστήρια. Θεωρώ πως τα δικαστήριά μας είναι ανεξάρτητα και δημοκρατικά. Εάν υπάρχουν στοιχεία που συνήθως είναι δίκαιε οι δίκε. Περνάμε τώρα στον εκπρόσωπο της Μάλτας, ο Γκαλέα. Buonasera al signor Galea, cinque minuti per la sua eh, presentazione. Prego. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Έχετε 10 λεπτά να κάνετε την παρουσίασή σας. Thank you, Mr. Ε, πέντε λεπτά σας ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή στη μητρική μου γλώσσα Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί με καλέσατε σήμερα εδώ να... Ε, σε σχέση με τον προτινόμενο διορισμό μου ως μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, όπως θα είδατε και στο βιογραφικό μου σημείωμα, ε, είμαι νομικός και πολιτικός ταυτόχρονα. Από τα ε, πολύ νεανικά μου, από τα πρώτα νεανικά μου χρόνια. Γεννήθηκα λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο, μια οικογένεια με νέα παιδιά, με, ε, σπούδασα μουσική και ε, μου αρέσουν ιδιαίτερα τα θέματα πολιτισμού και τεχνών και για τα τελευταία 13 χρόνια είμαι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο σε θέματα ε, κοινωνικού δικαίου και εργασιακού δικαίου στην νομική σχολή στο τμήμα Δημοσίου Δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου τη Μάλτα. Ταυτόχρονα είχα την ευκαιρία να εργαστώ σε υψηλέ βαθμίδε τη ε, κυβέρνηση στη χώρα μου όπου ε, έπαιξα άμυξο ρόλο σε θέματα πολιτικής και σε θέματα λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ήμουν πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μάλτας Ε, στην κοινή ε, κοινοβουλευτική επιτροπή. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχω μακρά θητεία ως μέλος του Κοινοβουλίου, ε, ως Υπουργός. Υπήρξε επίσης και, και, πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Μάλτας. Έχω αναλάβει πάρα πολλά καθήκοντα διάφορες φύσεως, κοινωνικής πολιτικής στο Υπουργείο Ιστορικών επίσης και Ιστορικών Υποθέσεων, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Υγείας και ε, ε, με τον τρόπο αυτό έχω αποκτήσει μεγάλη εμπειρία. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι είχα σημαντικές αρμοδιότητες για ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της Μάλτας. Και συνεργάστηκα με υψηλού εξηματούχου στον τομέα ε, τη ε, κατάρτιση του προπολογισμού, τη διεξαγωγή ε, σχεδίων και, και της σωστής τους εκτέλεσης σύμφωνα με τις βέλτιστες διαχειριστικές και διοικητικές αρχές έπαιξε σημαντικό ρόλο στην μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα στη Μάλτα, καθώς και επίσης και στον τομέα ε, των, της μεταρρύθμισης των συντάξεων. Ήμουν μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την ένταξη της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχα σημαντικό, έπαιξε σημαντικό ρόλο και σε θέματα κατάρτισης και του προπολογισμού, όπως σας είπα. Ήμουν επίσης ε, ε, πρόεδρος του Κοινοβουλίου ε, και είχα εξελέγει ομόφωνα. Έπαιξε σημαντικό ρόλο λοιπόν και στον τομέα ψήφισης νομοσχεδίων κτλ. Και επειδή το ελεκτικό συνέδριο στη χώρα μου ε, βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, πρέπει να σα πω ότι ήμουν υπεύθυνο για το θέμα αυτό ε, και όσον αφορά τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά και όσον αφορά τι δραστηριότητε ε, του συνήγορου του πολίτη. Όταν προτάθηκα λοιπόν για το αξίωμα αυτό, θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι θα μπορούσα να αξιοποιήσω την εμπειρία μου προς την κατεύθυνση αυτή. Κοιτάξτε, ο κόσμος μας ε, μεταβάλλεται ταχύτατα. Και ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, συνεχίζει στα αγγλικά ο μιλητής και πιστεύω ιδιαίτερα ότι η λογοδοσία λοιπόν σε αυτό τον ταχύως μεταβαλλόμενο κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντική για να είμαστε σίγουροι ότι ε, οι πολίτε αισθάνονται εμπιστοσύνη στους πολιτικούς θεσμούς. Νομίζω ότι η εμπειρία έδειξε παντού ότι δηλαδή έδειξε ότι παντού όπου δεν υπάρχει λογοδοσία δεν υπά... όπου δεν υπάρχει έλεγχος θα το πω διαφορετικά, όπου δεν υπάρχει έλεγχος δεν υπάρχει λογοδοσία και όπου, και όπου δεν υπάρχει λογοδοσία δεν υπάρχει έλεγχος ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν, αν λείπουν αυτά τα συστατικά, τότε πού βρίσκεται η δημοκρατία γι' αυτό πιστεύω ότι θα εργαστώ προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τις βάσεις της ε, νομιμότητας, εξασφαλίζοντας ότι η πολιτικοί οι κυβερνήσει, οι πολιτικοί θεσμοί όλοι είναι υπόλογοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ η κυρία Γιάλα. Σας ευχαριστούμε. Καλώς ορίσατε κύριε Γκαλέα στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να επιμείνω σε ορισμένα από τα θέματα τα οποία θίξατε κι εσείς. Βεβαίως δεν αναπτύξατε, θίξατε γιατί δεν είχατε χρόνο στη διάθεσή σας. Εσείς λοιπόν κατά κάποιο τρόπο είπατε ότι εξειδικεύεστε σε θέματα εργατικού δικαίου. Από ό,τι κατάλαβα αυτή είναι η εξειδικευσή σας. Θέλω λοιπόν να μας πείτε λίγο περισσότερα Μα είπατε βεβαίω ότι ε, ήσασταν μέλο του Εθνικού Κοινοβουλίου ε, και ήσασταν υπεύθυνο για διάφορε επιτροπέ και, σε επιτρο... και σε επίπεδο ε, δημοσιονομικού ελέγχου. Αλλά ρωτώ συγκεκριμένα. Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλεγχο, θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποια άλλη εμπειρία. Υπάρχει επίση και κάτι άλλο, μια αντίφαση που θέλω να μα ε, ξεκαθαρίσετε. Στι απαντήσει σα, και μάλιστα πρέπει να σα πω ότι εσεί ε, που έχετε και μακρά εμπειρία ω υπουργό απόλυτα νόμιμο βέβαια σε αυτό το θέμα, είπατε ότι η διαδικασία απαλλαγής εσείς ποτέ ε, στα καθήκοντά σας δεν ασχοληθήκατε με τη διαδικασία απαλλαγής. Όταν όμως μας στείλατε μία επιστολή για να μας εξηγήσετε ε, ότι δεν έχουν βάσει τα άρθρα τα οποία εμφανίστηκαν στον τύπο για τις δραστηριότητε. σας, όπου, ε, εντάξει, ο τύπο μα το ανέφερε, ε, ο τύπος ανέφερε ορισμένα τέτοια στοιχεία. Πάντως στη συνέχεια, στην απάντησή σας, αναφερθήκατε ε, σε έλεγχο οργανισμών υπό τον έλεγχό σας. Οπότε θέλω να μου ξεκαθαρίσετε αυτή την αντίφαση. Από τη μια λέτε δεν είχατε... Α, τε, ε, ότι εσείς δεν εμπλακήκατε σε θέματα απαλλαγή και από την άλλη λέτε ότι, εμπλακ, ότι, ε, ε ότι πραγματικά είχατε ασχοληθεί με τις δραστηριότητε. Και αυτό με, με οδηγεί στα άρθρα που εμφανίστηκαν στον τύπο αναφέρθηκε μία σύμβαση τεσσάρων δις για το πρόγραμμα κατάρτισης των εργαζομένων. Θέλω να μας εξηγήσετε τι ποσοστό των συμβάσεων αυτών αφορούσαν ε, τις δικές σας εκλογικές περιφέρειες. Δύο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα απαντήσω με τη σειρά. Στον τομέα του δημοσιονομικού ελέγχου υπάρχουν, ε, προβλέπονται διαφορετικές φάσεις. Εγώ ο, ως υπουργό με άλλους εκπροσώπους του Υπουργείου μου, ανώτατος υπαλλήλου, έπρεπε να διασφαλίσω την εγκυρότητα της, ε, του προγραμματισμού του οικονομικού της χώρας ε, και σε επίπεδο δημοσιονομικού θα έπρεπε να φροντίσω έτσι ώστε οι προβλέψεις να είναι ρεαλιστικές και να υφίστανται σταθερά μορφές ελέγχου να επαληθεύονται για να είναι λειτουργικές. Θα χρησιμοποιήσω αν θέλετε και μία μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιεί και το ελεγκτικό συνέδριο υπάρχει μία αντιπαράθεση αν θέλετε σε επίπεδο επιχειρημάτων ανάμεσα στο κάθε ενδιαφερόμενο Υπουργείο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το δικό μου Υπουργείο και το Υπουργείο Οικονομίας της χώρας. Σε αυτή την φάση συζητάμε τους στόχους, βλέπουμε αν οι στόχοι αυτοί είναι ρεαλιστικοί και προσπαθούμε να ορίσουμε τους αριθμούς τους οποίους ο καθένας έχει ανάγκη και στο τέλος αφού καταλήξουμε κάπου γίνεται μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο και εγώ πρέπει να παρουσιάσω τις προτάσεις αυτές στο Κοινοβούλιο, να τεκμηριώσω τις προτάσεις αυτές και ε, να δώσω τις απαιτούμενες εξηγήσεις. Και εφόσον έχω τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ξεκινάμε τη διαδικασία εφαρμογής σε επίπεδο εφαρμογής υπάρχουν διαφορετικά ελεγκτικά επίπεδα. Υπάρχει ο εσωτερικός ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου, υπάρχει επίσης και ένα κυβερνητικό σύστημα ε, εσωτερικού ελέγχου, διαρκές θα έλεγα. Μερικές φορές το σύστημα αυτό ασχολείται με συγκεκριμένους τομείς, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία σε συνεχή εξέλιξη, η οποία ελέγχει την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Και πάρα πολύ συχνά ε, ε, υπογραμμίζεται ε, ένα συγκεκριμένο τομέα έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με αυτό. Και μετά έρχεται αν θέλετε ε, το θέμα του ε, ελεγκτικού συνεδρίου το ελεγκτικό συνέδριο έρχεται σε μια ιστερότερη φάση έτσι ώστε να εξετάσει καταρχάς τη συμβατότητα μιας συγκεκριμένης δαπάνης με τις προβλέψεις οι οποίες είχαν κατατεθεί και εκ των υστέρων παρουσιάζεται μια έκθεση αξιολόγησης η οποία γίνεται αντικείμενο συζήτησης στο Κοινοβούλιο. Αυτές είναι όλες οι φάσεις αν θέλετε ε, του δημοσιονομικού ελέγχου. Για την απαλλαγή Ίσως δεν κατανόησα σωστά την ε, ερώτηση την οποία είχατε υποβάλει στο ερωτηματολόγιο. Δεν υπάρχει στο δικό μας σύστημα ε, μια συγκεκριμένη πράξη σαφώς καθορισμένη όπου ένας υπουργός ή ο πρόεδρος να καταθέτει μια τέτοια επιστολή απαλλαγής. Δεν είμαι εγώ ο οποίος ε, κλείνω την διαδικασία, δεν είμαι εγώ ο οποίος ε, ορίζω πότε οι εθνικές αρχές αποφασίζουν ότι πρέπει να κλείσουν οι διαδικασίες και ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι ε, κανόνες. Αν μέσω απαλλαγής θεωρείτε ε, το ότι εγώ κατά τη διάρκεια της 20 ετούς εμπειρίας την οποία έχω σαν υπουργός υπήρχε εξωτερικός έλεγχος ή έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο του τομέα του οικονομικού στον οποίο ήμουν εγώ υπεύθυνο, αυτό ναι. Υπήρχε πάντα αυτό το οποίο ονομάζουμε στη χώρα μου πιστοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης ή των συγκεκριμένων δαπανών και γενικά δεν υπήρχε καμία προϋπόθεση και κανένας περιορισμός και καμία υποσημείωση από πλευράς του ελεγκτικού συνεδρίου της Μάλτας. Βέβαια το να είναι κανένας υπεύθυνο ενός μεγάλου Υπουργείου, ενός Υπουργείου με ένα μεγάλο ε, προϋπολογισμό, είναι σαφές ότι αυτό προκαλεί ορισμένες ε, ε, ορισμένες παρατηρήσεις και διαφέρονται μερικές φορές κάποιες ατέλειες και κάποιες αδυναμίες. Αλλά δεν έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα σχετικά με απαλλαγή των υπηρεσιών για τις οποίες ήμουν εγώ υπεύθυνο. Τώρα, σχετικά με το άρθρο στο οποίο αναφερθήκατε. Δυστυχώς πρόκειται για ένα άρθρο το οποίο ε, περιλαμβάνει ισχυρισμούς εντελώς μα εντελώς αβάσιμους. Εγώ έχω απαντήσει με συγκεκριμένα επιχειρήματα και μπορώ να δώσω αν θέλετε την απάντηση αυτή τη γραπτή, αυτό το μνημόνιο που το απαντητικό το οποίο έχω ετοιμάσει θα το δώσω στον πρόεδρό σας και μπορείτε να το έχετε και εσείς στη διάθεσή σας. Θα σας εξηγήσω όμως το άρθρο αυτό αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις. Η μία από τις περιπτώσεις αυτές υποτίθεται ότι έγινε πριν 23 χρόνια. Είναι μια υπόθεση η οποία εξετάστηκε προσεκτικά από το Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο της Μάλτας. Και τα συμπεράσματα στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου δεν έχουν καμία αναφορά σε μένα. Δεν υπάρχει πουθενά το όνομά μου, δεν εμπλέκομαι σε τίποτα αναφέρεται σε ορισμένες διαδικαστικές αδυναμίες του προγράμματος αυτού, το οποίο ήταν ένα νέο πρόγραμμα και δεν είχε στη διάθεσή του το κατάλληλο προσωπικό για να το διαχειριστούν, αλλά το ελεγκτικό συνέδριο δεν βρήκε καμία απόδειξη, παρατήρηση ή ένδειξη η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί αρνητική για το πρόσωπό μου. Η συγκεκριμένη αυτή υπόθεση ελέγχθηκε επίσης και από μια άλλη ανεξάρτητη επιτροπή η οποία ονομάστηκε Επιτροπή Καταπολέμησης Φαινομένων Διαφθοράς, η οποία δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση και στην έκθεσή της η συγκεκριμένη αυτή προσωρινή επιτροπή είπε ότι δεν υπάρχει ίχνος στοιχείου το οποίο να υποδεικνύει την προσωπική μου εμπλοκή σε η αδίποτε παρατυπία ή διαδικασία διαφθοράς πρόκλησης διαφοράς. Λοιπόν, από αυτές τις πληροφορίες που σας έδειξα αποδεικνύεται ότι εγώ δεν ενεπλάκην σαν Υπουργός ποτέ στην καθημερινή διαχείριση αυτών των προγραμμάτων δεν επηρέασα ποτέ, δεν άσκησα τη διακριτική μου εξουσία, δεν ανέτρεψα η αδίποτε απόφαση προς το δικό μου προσωπικό συμφέρον, εγώ έκανα αυτό που κάνει κάθε υπουργό, εγώ υιοθέτησα τις γενικές κατευθύνσεις, την γενική στρατηγική, έλεγξα την στρατηγική αυτή και κλήθηκα να την εφαρμόσω και αυτό έκανα. Και όταν το ελεγκτικό συνέδριο έκανε παρατηρήσεις για κάποιες ατέλειες, και παρατυπίες. Αυτό το οποίο έκανα είναι ο υπεύθυνο ο, ο γενικός διευθυντής που ήταν ε, στην συγκεκριμένη θέση αρμοδιότητας ε, για τον τομέα της εργασίας εφάρμοσε όλες τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Και επανεξετάστηκε μετά από τις αλλαγές αυτές ε, η περίπτωση και το ελεγκτικό συνέδριο σε αυτή την περίπτωση, αν διαβάσετε την έκθεση προσεκτικά, δεν κάνει καμία μα καμία αναφορά στο πρόσωπό μου. Είπαμε αυτό ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια, ήταν η προσπάθεια δημιουργίας νέων επαγγελματικών ε, ε, σχολών κατάρτισης, πρόκειται για ένα εντελώς μηχανισμό και είναι αλήθεια ότι ένας τέτοιος μηχανισμός έχει ορισμένα προβλήματα στην διοικητική του αν θέλετε ε, δομή στην αρχή της λειτουργίας σου, άμα τη γεννήση του δηλαδή. Κατηγορηματικά λοιπόν επαναλαμβάνω ότι ουδέποτε προσωπικά ενεπλάκην στη σύναψη ή ουδήποτε συμβολέου και η ασδήποτε σύμβασης οι οποίες όλες υπεγράφησαν από στελέχη του Υπουργείου μου σύμφωνα με τους κανονισμούς οι οποίοι ήταν τότε ενισχύ. Και όταν μετά από τις μελέτες και τις έρευνες οι οποίες έγιναν ε, πράγματι βρέθηκαν ότι πράγματι είχαν παραβιαστεί κάποιοι κανονισμοί σχετικά με τις δημόσιες αυτές προμήθειες, απελήθη ο υπεύθυνο για τις προμήθειες αυτές και άλλοι υπάλληλοι πέρασαν από ε, διαδικασίες δικατικού ελέγχου. Τώρα, σχετικά με τα 4 εκατομμύρια στερλίνες Μάλτας. Ε, το 98% ήταν ε, μισθολογικό κόστος. Λοιπόν, ο ισχυρισμός αυτός είναι ένας ισχυρισμός ο οποίος ρίπτεται θα έλεγα εντελώς ανεύθυνα εις βάρος αθώων ανθρώπων. Όταν κάποιος είναι καλείται να πληρώσει κάποιους μισθούς ε, και το κάνει αυτό μάλιστα με διαφανή και ηλεκτρονικό τρόπο, δεν υπάρχει κανένα θέμα ε, απάτης. Τώρα σχετικά με τα ποσοστά δεν τίθεται θέμα απόδοσης ποσοστών σε ιαδήποτε. Δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο του λέει ο πρόεδρος. Και σίγουρα δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα η οποία να ξεπερνάει το 2%. Παρακαλώ να είστε πιο σύντομος από εδώ και πέρα γιατί δεν θα υπάρχει κανένας χρόνος για άλλους. Χατζημαρκάκης. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για το 100% που λάβατε από το Κοινοβούλιο, πράγματι. Βεβαίως ξέρετε πως έχετε να γεμίσετε το παπούτσια του κυρίου Μπονίτσι που ήταν ε, κορυφαία μορφή από τη Μάλτα και δεν ξέρω κατά πόσο να έχετε έρθει σε επαφή ε, μαζί του γιατί θα θέλαμε βέβαια να συνεχίσετε και εσείς το έργο του και θα ήθελα να γνωρίζω ποια σημασία δίνεται στην ε, πολιτική αξιολόγηση της εργασίας σας γιατί τελικά είστε πολιτικός και είπα πως χαίρομαι εγώ για το ότι μπορείτε να κάνετε πολιτική αξιολόγηση και άρα θα σας ρωτούσα Υπήρχε ένα πρόσφατο παράδειγμα της Ελλάδας όπου ο κρατικός δημοσιονομικός έλεγχος οδήγησε στην κρίση στην οποία βρισκόμαστε. Θεωρείτε λοιπόν πως έχει η υπηρεσία σας ρόλο παρέμβαση σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πολιτικό το ερώτημα, θέλω όμως να ακούσω την άποψή σας. Όχι. Όσον αφορά την συνεννόησή μου με τον ε, καθηγητή τον κύριο Μπονίτσι, πρώτα απ' όλα έρθει σε επαφή μαζί του όταν πληροφορήθηκα πως οι αρχές της Μάλτας κόπευαν να με προτείνουν για να συζητήσω μαζί του. Και είχε την καλοσύνη να με ενημερώσει, να μου παρουσιάσει το μηχανισμό του ελεγκτικού συνεδρίου και γνωρίζω πως ο κύριος καθηγητής, ο κύριος έχει κάνει καλή δουλειά και ελπίζω να μπορέσω να διδαχτώ από την εμπειρία του και να την ε, συνεχίσω κι εγώ. Όσον αφορά την πολιτική μου εμπειρία, όπως είπα, νομίζω πως... Ε, ποια ήταν η εμπειρία μου. Εγώ κοίταγα ζητήματα οικονομίας, ε, αποτελεσματικότητας από την πτυχή και τη σκοπιά κάποιο ο οποίος ήθελε να κάνει ό,τι καλύτερο για τη χώρα του. Και ακόμα και όταν κοίταγα ζητήματα νομιμότητας και κανονικότητας ήταν υπ' αυτή την πτυχή. Τώρα, στο ελεγκτικό συνέδριο, εάν με ορίσετε, θα έχω την δυνατότητα να κοιτάω, να εξέταζω τα διαστήματα από διαφορετική σκοπιά και είναι νομίζω σημαντικό κάποιος με πολιτική εμπειρία με ένα νομικό και ένα πολιτικό μυαλό που έχει βρεθεί σε αρκετές ε, καταστάσεις οποίες έπρεπε να δω ζητήματα συμμόρφωσης, ε, ορθής διαχείρισης, ε, κανονικότητας ή να μπορέσω να αντιληφθώ του το ποιε είναι οι συνέπειε πολύπλοκων κανονισμών. Γιατί τι ελέγχουμε τελικά, ελέγχουμε την διοίκηση. Ζητήματα διοίκησης λοιπόν και θεωρώ πως κάποιος με τη δική μου εμπειρία και προσόντα και ικανότητες είναι σε θέση να συνεισφέρει ε, στο ε, ελεκτικό συνέδριο για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε καλύτερα πώς θα ανταποκριθούμε στην αποστολή του συνεδρίου και να έχουμε και καλύτερη συνεργασία βεβαίως και με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Γκαλέα, γιατί ξεκαθαρίσατε ε, περισσότερο τα ζητήματα ε, στη σχέση με τις απαντήσεις που μας δώσατε. Ε, με ικανοποιεί αυτό το οποίο είπατε για το σχεδιασμό. Τώρα, πολύ σύντομα. Κατά τη γνώμη σας, ποιος τομέας δαπανών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και περισσότερο έλεγχο από το Ελεκτικό Συνέδριο. Δεύτερη ερώτηση. Οι κρατικές προμήθειες είναι ο υψηλότερος ε, τομέας κινδύνου ως προς τη διαφθορά. Μιλώ για τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορείτε να κάνετε για να παρεμποδίσετε και, ή, και ή να σταματήσετε αυτό το μηχανισμό διαφθοράς και απάτης στον τομέα των κρατικών προμηθειών και βεβαίω ανάλογα με τι αρμοδιότητε και, την, ε, και τι δυνατότητε που έχετε ω μέλο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Και μία δήλωση και όχι ερώτηση. Αναφερθήκατε στην αποτελεσματικότητα ε, και, και στην αποδοτικότητα και είπατε ότι ως μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου θα ασχοληθείτε με αυτές τις δύο έννοιες ε, με ιδιαίτερη προσοχή. Σας ενθαρρύνω, συμφωνώ απόλυτα. Βεβαίω θα πρέπει να αξιολογούμε τις, την, τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των ε, ε, σχεδίων που αποτελούν δικείμενο χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις ερωτήσεις σας. Κοιτάξτε, όσον αφορά τους ε, τομείς που θα, που θα απαιτήσουν περισσότερη προσοχή, τομείς του, του προπολογισμού, ναι, εκεί όπου ο κίνδυνος είναι υψηλότερο. Και και όπου ε, υπάρχει μεγαλύτερη επίδραση στις συνολικές ε, δηλώσεις αξιοπιστίας. Διότι φαίνεται από τις εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου ότι υπάρχει ε, μία κάποια βελτίωση σε ορισμένους τομείς. Ήδη δηλαδή έχουμε θετική γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά τους λογαριασμούς. Τους δημοσιονομικούς λογαριασμούς και τα αποτελέσματα. Επίσης υπάρχει βελτίωση στο επίπεδο νομιμότητας ε, σε αρκετούς τομείς. Αλλά κοιτάξτε, όταν εξετάσουμε ένα σημαντικό τομέα, όπως για παράδειγμα το τομέα συνοχής, εκεί υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Εγώ βεβαίω δεν είμαι ακόμα μέλος του ελεκτικού συνεδρίου ε, και ούτε υπήρξε στο παρελθόν, άρα θα πρέπει να διδαχθώ πολλά από τα ε, παλαιότερα μέλη του ηλεκτρικού συνεδρίου, αλλά γνωρίζω ότι το ηλεκτρικό συνέδριο ήδη ασχολείται με αυτούς τους ε, τομείς που παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει καλύτερους μηχανισμούς προς την κατεύθυνση αυτών των τομέων ιδιαίτερα. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όπου, ε, ότι, για το ότι το, το ελεκτικό συνέδριο προσπαθεί να κατανείμει καλύτερα τους πόρους του έτσι ώστε να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένους τομείς. Και προσπαθεί να πει, ε, να μεταφέρει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ε, το τι ακριβώς γίνεται σε αυτούς τους τομείς υψηλού κινδύνου και ε, τι θα μπορούσε να συστήσει. Και συμφωνώ μαζί σας ότι θέματα όπως για παράδειγμα κρατικών προμηθειών είναι ιδιαίτερα λεπτά και ευαίσθητα ζητήματα. Το γνωρίζω ότι ακόμα και στη χώρα μας μερικές φορές στις κρατικές προμήθειες προκύπτει η ανάγκη περαιτέρω εξασφάλιση ζητημάτων νομιμότητας. Για τις απάτες. Πολύ ευαίσθητος ε, τομέας και πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα κανείς θα πρέπει να διαβάσει τη συνθήκη. Και εκεί θα δει ότι η ευθύνη παρακολούθησης και δίωξης ε, θεμάτων ε, απατών και διαφθοράς ε, έγκυται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά τώρα και στα κράτη-μέλη. Το ελεκτικό συνέδριο πιστεύω ότι και εδώ μπορεί να παίξει ένα ρόλο για να εξασφαλίσει ότι κατά την άσκηση του ελέγχου υπάρχει απαραίτητη προσοχή και ο, ο επαγγελματισμός έτσι ώστε να δούμε το κατά πόσον τα σφάλματα αυτά είναι καθαρά σφάλματα ε, ή ε, σφάλματα εκ προθέσεως. Τότε, αν πρόκειται για πρόθεση, κανείς θα πρέπει να ε, προχωρήσει περισσότερο την έρευνα έτσι ώστε να εντοπιστούν σε πληρέστερο βαθμό οι τομεί που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτέ τι καταστάσει. Και τι μπορεί να κάνει το Ελληνικό Συνέδριο στη συνέχεια, είναι να παραπέμψει στην Όλαφ την υπόθεση και να υπάρξει κατάλληλη συνεργασία σύμφωνα με τι συνθήκε, με τι διατάξει συνθήκη. Ευχαριστώ, Γκρέσλερ. Ευχαριστώ. Ανησυχώ κάπως γιατί κάθε χρόνο κάνουμε αυτή τη συζήτηση με το Ελληνικό συνέδριο και δεν καταλήγουμε πουθενά. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν για να πάμε στην κατεύθυνση που ανέφερε ο κ. Χατζημαρκή. Χρειαζόμαστε κάποιε ουσιαστικέ βελτιώσει για το πώ δηλαδή καταρτίζονται οι εθνικοί λογαριασμοί και οι δηλώσει. Ε, και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Στην Ελλάδα πήγαμε και γνωρίζαμε πώ υπήρχε, εν περιπτώσει, μόνο εν μέρη λειτουργία του συστήματο των λογαριασμών. Το ξέραμε γιατί το ελληνικό κράτος ε, αποστέρισε από το ελληνικό ελεγκτικό συνέδριο τη δυνατότητα να κάνει σωστά τη δουλειά του. Οπότε πρέπει... Πού θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να δώσουμε βάρος και όσον αφορά και τα κονδύλια και την ε, χρηματοδότηση. Είναι πολύ ακαθόδες το ερώτημα. Τι σκοπεύετε να, να κάνετε. Είναι απάντηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Το ελεγκτικό συνέδριο οπωσδήποτε και υπό το φως των νέων διατάξεων. εξακολουθεί να παραμένει υπεύθυνο για τον έλεγχο της εφαρμογής του προπολογισμού, αλλά σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και είναι σαφή η συνθήκη πως τα κράτη-μέλη πρέπει να αρχίσουν να υπομίζονται μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά τη λογοδοσία, την διαβεβαίωση και πλέον οι συνθήκες τους ζητούν να συντονίσουν ε, τα εσωτερικά τους ε, συστήματα. Κατ' ουσίαν δηλαδή οι νέες συνθήκες λένε στα κράτη-μέλη σου λουποθείτε. Βεβαίως όλοι συμφωνούν επί της αρχής με κάτι τέτοιο. Και νομίζω πως το ελεγκτικό συνέδριο ήδη αναζητεί το πώς θα συνεργαστεί καλύτερα με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Γνωρίζω την ε, πολυπλοκότητα, έχουμε 27 κράτη-μέλη με 27 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Αντιλαμβάνομαι πως το ελεγκτικό συνέδριο έχει ξεκινήσει ένα κοινό πρόγραμμα ελέγχων με κάποιες χώρες και νομίζω πως αυτό αυτό θα μπορούσε να είναι το μέλλον, αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί εγώ το βρίσκω αδιανόητο, να έχουμε αυτή την κατάσταση, δηλαδή ένα κράτος μέλος να μην δίνει στο ελεγκτικό συνέδριο τους απαραίτητους πόρους για να λειτουργήσει. Σύμφωνα με το μαλτέζικο σύστημα, το ελεγκτικό συνέδριο έχει πολύ ισχυρή νομοθετική βάση, αποφασίζει μόνο του για τον προϋπολογισμό του, για τους πόρους του. Βεβαίω, εντάξει, γίνεται κάποια συζήτηση, αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει το ελεγκτικό συνέδριο. Αν θεωρεί πως χρειάζονται περισσότερους πόρους για να κάνουν αυτά τα οποία ορίζει το Σύνταγμα, μπορούν να τους ε, αποκτήσουν εξ λέγε, βάση του νόμου. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια κοινή τεχνική λύση, κοινές προδιαγραφές, έτσι ώστε τα διάφορα ελεγκτικά συνέδρια να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία τους γιατί βεβαίως ε, υπάρχει και η πρωτοκαθεδρία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αλλά πρέπει να σεβόμαστε την αυτονομία, την ανεξαρτησία των Εθνικών Ελεγκτικών Συνεδρίων. Αλλά σε, αυτή, τη, σε αυτόν τον αμοιβαίο σεβασμό νομίζω πως και το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να προχωρήσει σε αυτό το διάλογο μέσω της επιτροπές, των επιτροπών της επαφής που συνεδριάζουν τακτικά και γνωρίζω ήδη πως έχουμε αρκετές θετικές εξελίξεις από αυτές τις επιτροπές επαφής και από τους συνδέσμους με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό το οποίο ορίζουν οι συνθήκες. Γιατί αν τα κράτη-μέλη αναλάβουν την πραγματική ευθύνη για την ε, δήλωση για τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία διαχειρίζονται νομίζω πως ε, θα γίνει πιο αποτελεσματικό και το ελεγκτικό συνέδριο με το να επομίζονται και τα κράτη την ευθύνη. Οπότε μετά η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που θα επιβεβαιώνει την αξιοπιστία, την ε, αλήθεια των ε, εθνικών αυτών δηλώσεων θα μπορέσουμε και ως ελεγκτικό συνέδριο να διευκολύνουμε το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής σας δηλαδή, για να μπορέσετε και εσείς να ασκήσετε τα καθήκοντά σας ε, για να ελέγξετε και τα κρατημέλη και το Συμβουλίο. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκαλέα. Έρχεται ο κύριος Μπρόνισλαβ Κούμπιτς, προτινόμενος από την Πολωνία. Καλωσορίζω τον κύριο Κούμπιτ. Πέντε λεπτά έχετε για να κάνετε την παρουσίασή σα, κύριε Κούμπιτ. Κάτσε, να κάνω. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, είναι τιμή και ευχαρίστηση να βρίσκομαι για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ράτω με της ευκαιρίας να σας συστηθώ και να πω λίγα λόγια για την ε, μέχρι τώρα εμπειρία μου, καθώς και για τις προσδοκίες μου και τις ελπίδες μου όσον αφορά τα καθήκοντα που ελπίζω να αναλάβω στο ελεκτικό συνέδριο. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την σταδιοδρομία μου, να υπογραμμίσω πως όλη μου η σταδιοδρομία συνδέθηκε με τον έλεγχο, με την λογιστική και με τη διαχείριση της διοίκησης. Ως εσωτερικός έλεγκτης και επικεφαλής λογιστής ήμουν υπεύθυνο για τον εσωτερικό έλεγχο και για τα οικονομικά του ανθρακοριχείου στο οποίο εργάστηκα ως ε, διευθυντής της ΔΟΗ της Κατοβίτσε ήμουν υπεύθυνο για τα έσοδα και την διοίκηση βεβαίως της ΔΟΗ για τα οικονομικά της υπηρεσίας και για τον φορολογικό έλεγχο ως δε γενικός επιθεωρητής εσωτερικού ελέγχου είχα ιδιαίτερη ευθύνη για την εισαγωγή και τον συντονισμό και τη βελτίωση του εσωτερικού δημοσίου ελέγχου σε όλο τον δημόσιο τομέα της Πολωνίας. Ως σύμβουλος του Εθνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου ήμουν υπεύθυνο για την βελτίωση των εγγράφων που προετοίμαζε το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην τωρινή μου ιδιότητα είμαι υπεύθυνο για την πιστοποίηση δαπανών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης για το τμήμα οικονομικών αλλά και για την νομική υπηρεσία. Δηλαδή συνεργάζομαι με τις υπηρεσίες ελέγχου και με το Υπουργείο Οικονομικών. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω πως χάρη στην εμπειρία μου θα συνεισφέρω στις δραστηριότητες του ελεγκτικού συνεδρίου. Αλλά ελπίζω επίσης να κερδίσω και εγώ νέες εμπειρίες και να αντιμετωπίσω νέες προκλήσεις. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και τώρα είμαι έτοιμος να δεχτώ ερωτήσεις και ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιάλη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Κούμπικ ε, που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Κοιτάξτε, τώρα όσον αφορά τα επαγγελματικά σας προσόντα, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, γιατί τα, τα κάνατε όλα. Α, δεν ακούγατε. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίσατε κύριε Κούμπικ στην Επιτροπή μας. Η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνει η κυρία Γιάλα, ότι η απόψη επαγγελματικών προσόντων, πώς να το πω, γεννηθήκατε μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Και όσον αφορά τα δημοσιονομικά θέματα και θέματα ελέγχου. Τώρα, αυτή τη στιγμή ε, Ω Υπουργό τη Περιφερειακή Ανάπτυξη έχετε συγκεκριμένα καθήκοντα και μα είπατε ότι ακριβώ αυτό κάνετε. Πιστοποιείτε αυτά τα οποία αποτελούν αντικείμενο δημόσια συζήτηση και στην Επιτροπή μα. Το τμήμα συγχρηματοδότηση ε, εκ μέρου ε, των ε, εθνικών αρχών και των περιφερειακών. Είστε πρωταγωνίστε από ό,τι βλέπω τη περιφερειακή ανάπτυξη στην χώρα σα. Ακολουθώντα εν μέρει αυτό το οποίο έχουμε και εμεί στη χώρα μα στι αυτόνομε περιφέρειε. Λοιπόν, σα ρωτώ το εξή. Τρία πράγματα μάλλον τι λύση θα μπορούσατε να δώσετε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας ή μάλλον στα προβλήματα που δημιουργούνται όταν υπογράφουν ε, τις εθνικές δαπάνες Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας σε, στις περιπτώσεις της χρηματοδότησης. Τι λύση βλέπετε στα ομοσπονδιακά κράτη όπως η Γερμανία, στα ήμια ε, ε, ομοσπονδιακά όπως ε, η χώρα μου για παράδειγμα η Ισπανία. Εσείς επίσης επανειλημμένα αναφέρατε και βεβαίως αυτό είναι πολύ σωστό γιατί είναι ένα από τα κριτήρια τα οποία και εμείς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε για το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερα για το πώς βλέπετε το ζήτημα. Για το ελεκτικό συνέδριο προτείνει πολύ ενδιαφέρουσε πτυχέ προ την κατεύθυνση αυτή. Και τέλο. Στι απαντήσει σα βλέπω συνολικά κάποιο, ε, κάποιο στοιχείο περιπλοκότητα. Εσείς έχετε τόσα προσόντα και όσον αφορά τα θέματα δημοσιονομικά, τα φορολογικά, το ΦΠΑ, ε, μιλάτε κάπως περίπλοκα. Και όμως αυτό που μας ζητούν και τα κρατημέλη ε, και οι οργανώσεις ε, οι υπόλοιπε και εμείς οι ίδιοι ε, ζητούμε απλοποίηση όλων αυτών. Να γίνουν πιο απλά τα ζητήματα. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Πολωνία βρήκαμε μια λύση για, την, ε, για τις περιφέρειες στη χώρα μου και επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια. Ε, στην Πολωνία ε, ακολουθούμε κάποια επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία χωρίζουν σε δύο ομάδες. Πρώτα απ' όλα έχουμε τεχνικά προγράμματα και εδώ μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι, ε, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο και από την άλλη έχουμε τα προγράμματα τα οποία ε, ε, είναι περιφερειοποιημένα κατά κάποιο τρόπο. Στα πλαίσια των νέων προοπτικών εδόθη ένα μερίδιο στα, στις περιφέρειες και διαχειρίζεται με τον τρόπο αυτό και εκτελεί τα περισσότερα περιφερειακά προγράμματα η περιφέρεια. Αυτή είναι η απάντησή μου αν θέλετε. Όταν, θέλουμε δηλαδή να συμφιλιώσουμε το περιφερειακό επίπεδο με το εθνικό επίπεδο. Αυτή τη λύση ακολουθήσαμε την Πολωνία και ε, έδωσε καλά αποτελέσματα. Τα πρώτα βήματα αναλήφθηκαν ήδη σε επίπεδο των προηγούμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Και τώρα χρησιμοποιούμε την εμπειρία μας και εν ώψη των νέων προοπτικών δημιουργήσαμε 16 περιφερειακά προγράμματα. καθώς επίσης και ένα ευρύτερο πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συνοχής στην Ανατολική Πολωνία που είναι η περιοχή η λιγότερο αναπτυγμένη. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει πέντε περιφέρειες, ε, πέντε αυτόνομες περιφέρειες. Αυτό δείχνει ότι μπορούμε κάλλιστα να βρούμε μια επιχειρησιακή και λειτουργική λύση για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στο κεντρικό επίπεδο και στο περιφερειακό επίπεδο. Βεβαίω, με την ε, προπόθεση ότι ένα θα είναι ο αρμόδιο για το συντονισμό όλων αυτών των δράσεων. Και σε εμά αυτό ο συντονισμό ασκείται από το Υπουργείο Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παρά λοιπόν το, ε, την περιφερειοποίηση, έχουμε πετύχει τη συνοχή με τον τρόπο αυτό. Δεύτερη, στη δεύτερη σας ε, ερώτηση, όσον αφορά το ανεκτό επίπεδο κινδύνου και τα ασφάλματα. Και αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό, διότι συνδέεται άμεσα με το, ε, με το, με σύστημα εσωτερική διαχείριση. Για να μπορέσουμε τελικά να πετύχουμε την επίτευξη των στόχων μας. Με δύο λόγια μπορώ να σας πω ότι πρέπει να προσπαθούμε να πετύχουμε όσο να μεγαλύτερη ισορροπία στο συγκεκριμένο τομέα και να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στο κόστος ελέγχου και στα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών και τους στόχους που έχουμε ορίσει όσον αφορά τα αποτελέσματα. Κρατώντας βέβαια πάντα στο μυαλό μας το ε, επίπεδο, το ανεκτό επίπεδο ελέγχου που μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε. Αν δεχόμαστε μόνο ένα πολύ χαμηλό επίπεδο κινδύνου, τότε το κόστος ελέγχου ίσως ξεπερνά τα αποτελέσματα του ελέγχου. Βεβαίω υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναφέρεται στο ζήτημα αυτό και που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο συζητήσεων και προβληματισμού. Από το ίδιο το ηλεκτρικό συνέδριο. Ε, εγώ έχω διαβάσει ε, ε, προσεκτικά το έγγραφο και είδα ότι στο έγγραφο αυτό, όταν αναφέρεται το επίπεδο, το αποδεκτό επίπεδο ελέγχου, αυτό συνδέεται με το κόστος του ελέγχου και με τα αποτελέσματα, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά την απλοποίηση. Ο στόχο τη της μέγιστη απλοποίηση όλων των προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότηση από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Στόχο λοιπόν όλων των πολιτικών είναι η απλοποίηση, η απλούστευση έτσι ώστε να πετύχουμε το ελάχιστο δυνατό αριθμό ε, εσφαλμάτων. Όλες οι αναλύσεις ε, αποδεικνύουν ότι όσο πιο ε, περίπλοκο είναι το σύστημα, τόσο αυξάνεται το, το επίπεδο εσωτερικού κινδύνου. Άρα τελικά έχουμε αύξηση του κόστους του προγράμματος. Θα μπορούσα βεβαίως ε, να επεκταθώ πολύ περισσότερο ε, στο ζήτημα αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Ευχαριστώ. Κυρία Γιάλα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, σε σχέση με, τη, με την πρώτη σας ερώτηση. Εσείς ε, ασχολείστε με την εθνική πιστοποίηση, εθνική επαλήθευση των προγραμμάτων και του εθνικού και του προγράμματος για την Ανατολική Πολωνία, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεύτερον, εσείς είσαστε ελεκτής σε επαγγελματικό επίπεδο, θα εξακολουθήσετε να ασκείτε τη δραστηριότητά σας αυτή ή όταν ε, διοριστείτε ως μέλος του ελεκτικού συνεδρίου όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με το ζήτημα αυτό δεν θα τα θα, θα αφήσετε στην άκρη και δεν θα ασχοληθείτε πλέον. Ευχαριστώ. Odpowiem na pytanie pierwsze. Tak, osobiście jestem odpowiedzialny w imieniu... Πράγματι είναι θετική απάντησή μου. Εγώ θεωρώ ότι είμαι προσωπικά υπεύθυνο για την πιστοποίηση όλων των δαπανών που ε, αφορούν ε, είτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα εθνικά προγράμματα στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, όπως επίσης και τα περιφερειακά λεγόμενα προγράμματα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή η οποία έχει προταθεί για τις περιφέρειες και η οποία έχει ως εξής. Σε κάθε περιφέρεια υπάρχει μια υπηρεσία ή μια θηγατρική αν θέλετε υπηρεσία αυτής της υπηρεσίας πιστοποίησης. Και αυτή η θηγατρική υπηρεσία προχωρά στην ανεξάρτητη πιστοποίηση των δαπανών στα πλαίσια των περιφερειακών προγραμμάτων. Ακόμα όμως και αν υπάρχουν αυτές οι θηγατρικές, εγώ εξακολουθώ να είμαι υπεύθυνο για, για τον έλεγχο όλων των ε, εγγράφων τα οποία κατατίθεται και εγώ είμαι αυτός ο οποίος υπογράφει την πιστοποίηση στην τελική φάση. Είμαι και εσωτερικός και εξωτερικός ελεγκτής θα έλεγα δημοσιονομικός. Τι εννοώ με αυτό. Εγώ δεν ασχολούμαι με την εξωτερική μορφή ελέγχου εδώ και αρκετό καιρό και δεν ασχολούμαι επίσης και με την πιστοποίηση CAA δηλαδή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ισχύσει και στο μέλλον. Συνεπώς δεν υπάρχει εν πάση περιπτώσει κανένα θέμα σύγκρουσης ε, συμφερόντων. Μακοβέη, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Κούμπικ. Το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξής. Ε, ήσασταν, είστε τώρα στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ασχολείστε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε το ερώτημά μου είναι ποια συγκεκριμένα βήματα έχετε αναλάβει για την καταπολέμηση της απάτης. Αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ε, κάποια παραδείγματα και το τι σημασία θα έχουν στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεύτερο ερώτημα, όπως είπαμε και με τον προηγούμενο υποψήφιο, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ανασκουμποθούν μέσω και του Εθνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αλλά πώς θα αντιδράσετε, τι θα κάνετε αν αντιμετωπίσετε ένα Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο που δεν ε, θέλει να εκπληρώσει αυτά τα καθήκοντα. Ευχαριστώ. Για την πρώτη σας ερώτηση, στα πλαίσια των εσωτερικών διαδικασιών, έχουμε συγκεκριμένες, συγκεκριμένες μορφές ελέγχου, πολύ συγκεκριμένες, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντίστοιχες. Αν υπάρχει μία υποψία ή αν έχουν ήδη εντοπιστεί κάποιες περιπτώσεις απάτης ή κάποιες ε, περιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν ποινικέ κυρώσεις, τότε ενημερώνουμε αμέσως τα αρμόδια όργανα. Το σύστημα αυτό λοιπόν λειτουργεί στην Πολωνία. Έχουμε ένα σύστημα όπως είπα εσωτερικής ενημέρωσης, το οποίο λειτουργεί ως εξής. Η διαδικασία την οποία ακολουθούμε μεταφέρει τις, μετα, μεταφέρει τις πληροφορίες στη συγκεκριμένη υπηρεσία που ασχολείται ε, με τις ελεγκτικές διαδικασίες. Αυτή η υπηρεσία είναι ανεξάρτητη και είναι η υπηρεσία η οποία ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και όχι στο αρχικό Υπουργείο. Η υπηρεσία αυτή συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα και τα αποστέλει σε μια υπηρεσία α, ομόλογη θα έλεγα της ΟΛΑΦ. Αυτή η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει έναν υπεύθυνο κυβερνητικό υπάλληλο που ασχολείται με τις συγκεκριμένες μορφές απάτης όπως αυτή που στη συγκεκριμένη περίπτωση εντοπίζεται. τεκμηριώνει τις καταγγελίες οι οποίες υπάρχουν και όπως είπα τις επεξεργάζεται τις πληροφορίες αυτές η ΟΛΑΦ. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η συνεργασία ανάμεσα στο ελεγκτικό συνέδριο και τα εθνικά συστήματα ελέγχου, έτσι όπως λειτουργούν στην Πολωνία. Αντίστοιχα συστήματα υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Καταρχάς έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε επίπεδο συνθήκων. Οι τελευταίες εμπειρίες ε, από τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι τα πράγματα ε, συνεχίζουν να βελτιώνονται. οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ε, έχουν δίνει την συνεργασία τους ε, με το ελεγκτικό συνέδριο και αυτή η βελτιωμένη συνεργασία θα έλεγα βοηθάει πάρα πολύ τα πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, έτσι ώστε τα Εθνικά Κοινοβούλια να είναι σε θέση να πείσουν τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές που ασχολούνται με τις ελεγκτικές διαδικασίες και τα Εθνικά Κοινοβούλια να προτείνουν στο να συμπεριληφθεί στα πλαίσια του ελέγχου του κεντρικού οργάνου και η τομέα της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Στα πλαίσια του ελεγκτικού κεντρικού συνεδρίου εμείς δεν αρκούμεθα μόνο στον έλεγχο ε, που μας ζητείτε να κάνουμε σε συγκεκριμένες παραγγελίες, θα έλεγα, της Πολωνικής Βουλής ή των Πολωνικών Υπουργείων, αλλά ε, θα πρέπει να ελέγξουμε και τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται χρήματα που προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό σε αιτήσια βάση το κάνουμε αυτό, σε συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο του Λουξεμβούργου, επί τη βάση των προγραμμάτων τα οποία έχουμε αποφασίσει στο παρελθόν από κοινού. Αυτό πρέπει να γίνεται σεβόμενη βέβαια την ανεξαρτησία όλων των εμπλεκομένων οργάνων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσετε λίγο τις προθεσμίες οι οποίες μεσολαβούν για τη χορήγηση της απαλλαγής. Γίνονται εδώ και 20 χρόνια προσπάθειες, λέει ο κ. Σόντι, για την συντόμευση αυτής της περίοδου και προσπαθούμε να επιταχύνουμε κάπως τα πράγματα. Και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Μας δίδονται οι λογαριασμοί τον Ιούλιο σαν παράδειγμα, το ελεγκτικό συνέδριο μας δίδει τη γνωμοδότησή της τον Οκτώβριο του επόμενου χρόνου και έχουμε έξι μήνες κανονικά για να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο που απαιτείται και να ψηφίσουμε τον επόμενο Απρίλιο. Μήπως θα μπορούσαμε να συντομεύσουμε τη διαδικασία αυτή κατά ένα τρίμηνο Έτσι γίνεται σε πάρα πολλές χώρες, όπως τη συγκεκριμένη από την οποία προέρχομαι. Ε, μπορούμε να έχουμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου στο δεύτερο τρίμηνο του επομένου χρόνου, έτσι ώστε να έχουμε ένα εξάμηνο και στο τέλος της χρονιάς να μπορέσουμε να κλείσουμε δηλαδή λιγότερο από ένα χρόνο μετά τους λογαριασμούς και να χορηγήσουμε ή όχι την απαλλαγή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το θέμα ε, το οποίο θέσατε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και απαιτείται να υπάρξουν ορισμένες αποφάσεις ε, το ταχύτερο δυνατόν. Από την άλλη είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιταχύνουμε κάποιες διαδικασίες, ιδιαίτερα όταν έχει μάθει το σύστημα να λειτουργεί με συγκεκριμένους ρυθμούς για πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να σας ε, μεταφέρω μια εμπεριστατωμένη άποψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ε, δεν ελέγχω σε τέτοιο επίπεδο λεπτομέρειας ε, το χρονισμό θα έλεγα και δεν μπορώ να γνωρίζω τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για κάθε όργανο έτσι ώστε να επεξεργαθεί τα στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στη χορήγηση της απαλλαγής το σύστημα δαπανών σαν παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι περίπλοκος και είναι πολύ δύσκολο να δώσω μια σαφή απάντηση. Είναι σαφές βέβαια ότι θα πρέπει να συντομευθούν οι διαδικασίες, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους μπορούμε να κάνουμε βήματα σμίκρινσης του χρόνου που απαιτείται εμείς δεν θέλουμε βέβαια σε καμία περίπτωση να υπάρξει ε, μια συνέπεια από την συντόμευση των διαδικασιών, συνέπεια αρνητική για την ποιότητα του ελέγχου. Αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Πάντως μπορεί να γίνει μια ανάλυση σε βάθος της δημοσιονομικής διαδικασίας εξ εξ των υστέρων. Έχουν ξεκινήσει κάποιες πρώτες σκέψεις στο ελεγκτικό συνέδριο και οι αναλύσεις αυτές θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα τα οποία θα προταθούν σε υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα σε λίγο καιρό. Τώρα αν τα συμπεράσματα αυτά πράγματι θα επιτρέψουν να διορθωθεί η κατάσταση δεν μπορούμε να ξέρουμε. Είναι κάτι το οποίο θα φανεί στο άμεσο μέλλον. Πάντως θα πρέπει από κοινού να δώσουμε μια απάντηση που να μειώνει τον χρόνο. Κλείνοντας να πω ε, ένα πράγμα μόνο γιατί όπως σημειώσατε στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν έδωσα συγκεκριμένη απάντηση. Η διαδικασία απαλλαγής είναι μια βαριά διαδικασία, είναι μια διαδικασία ε, ιδιαίτερος περίπλοκη. Υπάρχουν διαδοχικές εκθέσεις οι οποίες παρουσιάζονται από διάφορες υπηρεσίες για να κριθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Υπάρχει η DAS, η δήλωση αξιοπιστίας, υπάρχουν επίσης ε, και οι μορφές ελέγχου απόδοσης ή επίδοσης μάλλον, ε, το performance audit. Υπάρχουν λοιπόν παράλληλες πολλαπλές διαδικασίες, πρέπει ταυτόχρονα να δοθεί η δυνατότητα στις υπηρεσίες ή στα όργανα τα οποία καταλογίζεται κάτι να εκθέσουν τα επιχειρήματά τους και μετά από το peer review το οποίο γίνεται σε επίπεδο του ελεγκτικού συνεδρίου το πρώτο στάδιο ανάλυσης τότε μόνο θα έχουμε μια δυνατότητα απάντησης. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας θα ακούσουμε τον Σλοβάκο υποψήφιο, τον κύριο Μπάλκο. Καλωσορίζω τον κύριο Μπάλκο, έχει πέντε λεπτά. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Συγγήτρια, κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές, είναι τιμή και ευκαιρία που έχω σήμερα την δυνατότητα να σας συστηθώ ως προσήφιος για μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Για να μην διαβάζετε το βιογραφικό μου θα ήθελα να σας συστηθώ μέσω της δηλωσής μου. Ήρθα με αρκετή ταπεινότητα εδώ πέρα γιατί βλέπω πως Έχουμε εδώ πέρα πρώην ευρωβουλευτές, ε, βουλευτές ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια, πρώην υπουργού, ε, εκπροσώπους των διαφόρων κομμάτων και ειδικού στα νομικά, τα λογιστικά κτλ. Βεβαίω έχουν μια εμπειρία για τη λειτουργία των δημοσίων αργών στο εθνικό, το διεθνές και το τοπικό επίπεδο. Βεβαίως ε, ξέρουμε πως οποιαδήποτε δημόσια αρχή για να υπηρετήσει τους πολίτες από τους οποίους ε, αντλεί τη δυναμή της ε, πρέπει να έχει και τους απαραίτητους πόρους. Και εσείς, η Επιτροπή σας φροντίζεται να χρησιμοποιούνται σωστά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, υποψήφιο μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα ήθελα και εγώ και θα ήμουν περήφανος να σας βοηθήσω στα καθήκοντά σας. Βεβαίως κάθε υποψήφιος που έρχεται ενώπιον της Επιτροπής σας θα ε, ήθελε να σας πείσει πως η δική του συνεισφορά θα βοηθήσει την εφαρμογή του κοινοτικού προπολογισμού. Ελπίζω λοιπόν η ακρόαση αυτή και η ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε θα αποτελέσουν την αρχή μιας καλής συνεργασίας και επιτυχούς συνεργασίας. Έχω εμπειρία δύο δεκαετιών στα δημόσια οικονομικά σε τρεις Πρώτα απ' όλα είχα διάφορες διοικητικές θέσεις στον τραπεζικό τομέα. Δεύτερον, έχω διοικητική εμπειρία στη δημόσια διοίκηση. Τρίτον, ε, θεωρώ ένα θετικό σημείο το ότι ήμουν ε, αναπληρωτής καθηγητής στον τομέα του δικαίου των οικονομικών και βεβαίως είχα συμμετάσχει και στην σύνταξη ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης. Γνωρίζω το ότι ο προϋπολογισμός και τα δημόσια οικονομικά δεν αφορούν μόνο τα έσοδα και τα έσοδα και τους αριθμούς, αφορούν και τις πολιτικές αξίες και τους στόχους τους οποίους εκφράζεται ως εκπρόσωποι των διαφόρων πολιτικών ομάδων και το σημαντικότερο ως ερετή εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Οπότε έχουμε και την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη θέση ενισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας, ειδικά όσον αφορά την διαδικασία του προϋπολογισμού. Οπότε μπορούμε να κατευθύνουμε και τις επενδύσεις και να καθορίσουμε τον προπολογισμό, πράγματα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά και εδώ θεωρώ πως παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ο έλεγχος μέσω του ελεγκτικού συνεδρίου. Με την εμπειρία που αποκτήσαμε από την οικονομική κρίση πρέπει να διασφαλίσουμε πως το κάθε ευρώ ξοδεύεται με τον καλύτερο τρόπο. Ως ε, μέλος του Κοινοβουλίου θα ήθελα και εγώ να σας βοηθήσω για την διαχείριση αυτού του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συγγήτρια, κύριε και με τις πρώτες αυτές αγωγικές παρατηρήσεις ε, ανέφερα κάποιες από τις ιδέες μου όσον αφορά τις δραστηριότητε μου ως μελλοντικό μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπάρχουν και άλλες ιδέες που έχω αναφέρει στις γραπτές μου απαντήσεις. Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα προσπαθήσω να απαντήσω τις ερωτήσεις σας, ελπίζω ικανοποιητικά και αν μου επιτρέπετε τώρα θα συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα. Δεδομένου δε του ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα μου στην Επιτροπή σου ακουστεί εδώ πέρα για πρώτη φορά. Και τώρα είμαι διατεθειμένος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Στο κυρία Γιάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μπάλκο. Στην επιστολή που μας στείλατε, οι απαντήσεις ε, στις ερωτήσεις μας με κάνουν να πιστεύω πως ε, θα απαντούσατε σε διαφορετικές γλώσσες και όχι μόνο στα αγγλικά. Οπότε χαίρομαι για το ότι χρησιμοποιήσετε και τη δική σας γλώσσα. Με βάση την εμπειρία σας, ε, την εμπειρία σας στον τραπεζικό τομέα κτλ. Και ήσασταν βεβαίως και πανεπιστημιακός ε, δάσκαλος και τώρα είστε σύμβουλος του Πρωθυπουργού και συχνά συναντάτε τους φοιτητέ σας στη δημόσια διοίκηση, σε τράπεζες, σε ελεγκτικούς φορείς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σκοπεύετε να κάνετε Παραδείγματο χάρη, ναι, αν γίνετε μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, τι σκοπεύετε να κάνετε εάν δεν ε, συμφωνήσετε με π.χ. τον Πρωθυπουργό σας ή έναν από τους πρώην φοιτητές σας. Γιατί είναι και δύσκολο να τους επιπλήξετε. Επίσης, η απάντησή σας στην ερώτηση του τι θα κάνετε εάν ε, το Κοινοβούλιο αποφασίσει πως δεν είστε ο καταλληλότερος για αυτή τη δουλειά, δεν ήταν και πολύ σαφής. Η απάντησή σας ήταν κάπως ε, αμφίσιμη. Και κάτι άλλο που με ανησύχησε ήταν το πώς βλέπετε τις δραστηριότητες σας σε σχέση με την Επιτροπή. Είπατε πως ε, ένα μέλος του γραφείου σας θα ασχολείται με την Επιτροπή μας. Εμείς ελπίζαμε πως ο ίδιος εσείς προσωπικά θα ε, ήσασταν σε επαφή μαζί μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, επέλεξα την Σλοβακική γιατί γνωρίζω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει και την πολυγλωσία και ευχαριστώ μιλάω σλοβακικά γιατί δεν υπάρχει και σλοβάκος ε, βουλευτής στην Επιτροπή σας και καλό θα είναι κάποιοι να ακούσουν τουλάχιστον και έστω και μία φορά σλοβακικά. Τώρα για το τι θα κάνω εάν δεν με υποστηρίξετε. Ε, εντάξει, η διαδικασία προβλέπει πως η εθνική κυβέρνηση πρέπει να ε, συμφωνήσει, οπότε θα συντονιστώ με την Σλοβακική κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό, τον ε, Αντιπρόεδρο της ε, κυβερνήσεως, αλλά βεβαίως από ηθική σκοπιά καλό θα ήταν να αποσύρω την υποψηφιότητά μου γιατί η συνεργασία μου μαζί σας είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να είμαι το μακρύ χέρι της Επιτροπής σας. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει 800 υπαλλήλους και η Επιτροπή σας δεν έχει και τις τεχνικές δυνατότητες ε, για ούτε καν ε, το προσωπικό αυτό. Οπότε πρέπει να συνεργαστούμε πάρα πολύ στενά, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα ακριβώς ένα από τα ερωτήματά σας, γιατί σκεφτόμουν ήδη την απάντησή μου. Μπορείτε λοιπόν να επαναλάβετε το τελευταίο ερώτημά σας. Κοιτάξτε, η τελευταία ερώτηση ήταν η εξή. Εσεί στι απαντήσει σα μιλήσατε για τη σχέση με την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Κοινοβουλίου και για το γεγονό ότι θα, θα ορίσετε ένα μέλος του γραφείου σας για την παρακολούθηση. Αλλά εμείς θέλαμε εσείς ο ίδιος. Δεν απαντήσατε όμως για την ανεξαρτησία. Δηλαδή, ε, όταν υπάρχει ε, πρόβλημα με τον ε, Πρωθυπουργό σας ή μερικές φορές και με τους μαθητές σας. Ναι, πράγματι. Το, το πιο απλό είναι το τελευταίο ερώτημα. Πώς βλέπω τη συνεργασία. Πράγματι είχα σκεφτεί. Εννοώ ότι ένα άτομο θα ασχολείται καθημερινά με αυτή τη δουλειά και θα με ενημερώνει. Βεβαίως η επαφή μας δεν θα γίνεται μόνο μέσω ενός συνεργάτη μου, θα έχετε προσωπική επαφή ε, μαζί μου, σε σημείο που θα είναι ίσως και δυσάρεστο, γιατί θα με βλέπετε τόσο συχνά και θα ακούτε τις προτάσεις και τις ιδέες μου όσον αφορά τώρα την ε, ανεξαρτησία. Ε, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα εγώ να είμαι απέναντι από τους πρώην μου ή τις ε, εθνικές ε, αρχές. Νομίζω ολόκληρη η προσωπική μου διαδρομή συνδέεται με τα δημόσια οικονομικά και πάντα εγώ προσπαθούσα να προστατεύω τα, χρή... τα χρήματα των φορολογουμένων και αυτό δίδασκα και στους φοιτητές μου. Ε, είδα και εγώ και τα δικά σας βιογραφικά σημειώματα. Γνωρίζω πως εσείς είστε νομικός και όχι μόνο γλωσσομαθείς, οπότε αντιλαμβάνομαι πως ε, το δίκαιο το σχετικό με τα οικονομικά δεν ήταν πάρα πολύ ελκυστικό και προσπάθησα να εξηγήσω πως η προστασία των δημοσίων συμφερόντων ε, μπορεί να προσφέρει πολλές ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Και ευχαρίστως ε, να προωθήσω και το έργο της Επιτροπής σας, γιατί πολλοί υπουργοί και υφυπουργοί με ρωτάνε τι είναι ακριβώς αυτό το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν είναι γνωστό ότι είναι ένα από τα πέντε βασικά θεσμικά όργανα της ε, Ένωσης και η καθημερινή του δουλειά είναι να προστατεύει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Οι ριαλάζουν αλλάζουν, οι απόψεις ε, αλλάζουν. Γι' αυτό θα ήθελα και εγώ στη μελλοντική μου εργασία να ανυψώσω την προστασία των δημοσίων οικονομικών και στην χώρα μου σε ένα υψηλότερο επίπεδο και να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το ελεγκτικό συνέδριο στην χώρα μου και βεβαίως ε, θα ενημερώσω και για το έργο της δικής σας επιτροπής. Σα Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε κύριε Μπάλκο. Έχω δύο ερωτήσεις στη χώρα σας ασχοληθήκατε με μέτρα που αφορούσαν την εισαγωγή του ευρώ στη Σλοβακία. Το ερώτημα είναι το εξής. Πώς αξιολογείτε τη μεθοδολογία ε, για την υποβολή μακροοικονομικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και στα άλλα, ε, και στα, και στα άλλα ευρωπαϊκά, στους άλλους ευρωπαϊκούς ευρωπαϊκού οργανισμού. και γιατί σας το λέω αυτό, γιατί έχω στο μυαλό μου την πρόσφατη περίπτωση της Ελλάδας και την υποβολή των στοιχείων. Δεύτερον, θα αλλάζατε την αξιολόγηση του αριθμού των σφαλμάτων ε, σε σχέση με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ρωτώ αυτό, διότι ο μέσος όρος που έχουμε για, τους, τις 27 χώρες μέλη ε, είναι αυτό που είναι, αλλά δεν νομίζουμε ότι ο μέσο όρο είναι σχετικό, είναι σημαντικό, γιατί υπάρχουν μεγάλε διαφορέ ε, ανάμεσα στο, ε, στο ανώτατο όριο και στο κατώτερο. Γι' αυτό θέλουμε την άποψή σα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να δούμε ε, τα στοιχεία σε κάθε κράτο μέλο ή να αναφερόμαστε στον μέσο όρο. Ευχαριστώ. Ε, ναι. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ερώτημά σας. Τα νούμερα είναι πάντα έτσι λίγο παραπλανητικά. Προσωπικά αντιλαμβάνομαι πως ε, τα στατιστικά στοιχεία αφορούν βεβαίως ε, και τους ε, μέσους όρους, αλλά πρέπει να υπάρχει εξειδικεύση ένα κράτος μέλος, π.χ. Αυστρία, Γερμανία και Φιλανδία όσον αφορά την οικονομική πολιτική έχουν ε, ποσοστό σφάλματος μικρότερο από 1% και Ρουμανία, Βουλγαρία έχουν ποσοστό σφάλματος πάνω από 13% και ο μέσος όρος μετά είναι κάπου στη μέση. Θεωρώ λοιπόν πως ε, πρέπει να κάνουμε τα πράγματα ως ε, εξής. Ε, το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης ή το ΑΕΠ κατά κεφαλή να αποτελέσει ένα κριτήριο. Νομίζω ότι είναι καλύτερο κριτήριο. Και τώρα όσον αφορά τη μεθοδολογία για την εισαγωγή του ευρώ. Στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή σας, έχει ακουστεί πολλές φορές έχει υποθεί πως ε, μήπως οι χώρες με μικρότερη οικονομική ανάπτυξη θα έπρεπε να έχουν πιο ήπια κριτήρια από αυτές που είναι πιο ανεπτυγμένες. Εγώ θεωρώ πως ε, τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν, τα πέντε κριτήρια ε, ή τα τέσσερα κριτήρια σύγκλησης είναι σωστά, είναι αρκετά ρεαλιστικά και είμαι πεπισμένος πως ε, έχουν επιλεγεί σωστά τα κριτήρια, παραδείγματος χάρη. Το έλλειμμα του ΑΕΠ 3% ε, δεν είναι ενιαίο κριτήριο καμία χώρα ή, ή παραδείγματος χάνει το 60% ποσοστό του δημοσίου χρέους. Βεβαίως σήμερα έχουμε μέχρι και 100% χρέος. Αλλά αυτό δεν θα διαρκέσει για πάντα. Θα έλεγα πως είναι μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης να μην πω πολέμου. Αλλά... Πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε αυτά τα κριτήρια. Ε, είχαμε και ε, φόβο βέβαια στην Σλοβακία για τα, τα αυτά. Εγώ όμω είμαι πεπισμένο πως είναι σωστά και εφαρμόζονται σωστά. Αν δεν υπάρχουν... Α, έχετε να ρωτήσετε κάτι. Να πω δύο λόγια. Να πείτε δύο λόγια μάλλον, αν ε, μπορείτε, για τη μεθοδολογία υποβολή στοιχείων. Θα αλλάζετε κάτι στο θέμα αυτό. Neviem, ξέρω τώρα σε ποια μεθοδολογία ακριβώς αναφέρεστε. Μιλάτε για το έτος αναφοράς. Όταν θέλει μια χώρα να ενταχθεί στο ευρώ. Σύμφωνα με την εμπειρία μου, μπορώ να πω πως η μεθοδολογία στην περίπτωση της Σλοβακίας δεν ε, δημιούργησε προβλήματα. Οπότε βασίζομαι τώρα στη δική μας ε, εθνική εμπειρία. Μια χαρά ήταν η μεθοδολογία και εφαρμόστηκε στην ε, Σλοβακία. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπάλκο και να καλέσουμε τον επόμενο υποψήφιο των Ιρλανδικών Αρχών, τον κύριο Έωιν Οσί. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σι. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εξέτοιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη τιμή βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας δεχόμενο την υποψηφιότητα από την κυβέρνησή μου ε, ω υποψήφιο μέλο του ε, Ελεκτικού Συνεδρίου. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα ενώπιον τη Επιτροπή σα, διότι πιστεύω ότι κάθε μέλο του Ελεκτικού Συνεδρίου χρειάζεται μια συγκεκριμένη εντολή από του ε, άμεσα εκλεγμένου ε, ευρωβουλευτέ που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των φορολογουμένων τη Ευρώπη. Αν εγκρίνετε την υποψηφιότητά μου, με μεγάλη μου χαρά θα ε, θα εξακολουθήσω να είμαι, ε, ε, να, θα, θα, να είμαι ως μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου για τα υπόλοιπα δύο χρόνια. η κυρία Γκέγεν Κουίν τώρα έγινε μέλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν συμφωνείτε τα υπόλοιπα δύο χρόνια, τα υπόλοιπα δύο χρόνια θα πάρω εγώ τη θέση της. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Τα, νομίζω ότι τα προσόντα μου φαίνονται μέσα από, την, από τις απαντήσεις της ερωτήσεις που μου θέσατε θα ήθελα να τονίσω, να, να δώσω έμφαση σε ορισμένα σημεία, τα οποία νομίζω θα σας βοηθήσουν όταν θα πάρετε την απόφασή σας. Είμαι μέλος του Συμβουλίου των Ορκωτών Λογιστών στην Ιρλανδία. Τα μέλη του Ινστιτούτου με εξέλεξαν για να τους εκπροσωπήσω ε, στο Συμβούλιο τους που είναι το, ε, ε, το όργανο, το διαχειριστικό όργανο του, του κλάδου στην Ιρλανδία. Εργάστηκα ως ορκωτής λογιστής, ε, είμαι σύμβουλος ε, ε, σε φορολογικά ζητήματα, έχω τον τίτλο του δικηγόρου, έχω σημαντική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, στον τομέα των επιχειρήσεων και αυτό το οποίο παρουσιάζει ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον για σας είναι η συμμετοχή μου στην, στα λογιστικά της κυβέρνησης. Ήμουν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Αστυνομίας της Ιρλανδίας πρόκειται για σημαντική θέση, διότι διότι πρόκειται για συμβουλευτικό έργο προς τον Διευθυντή της Αστυνομία για τη δαπάνη του 1,5 δις ευρώ το χρόνο. Επίσης, με διόρισε η κυβέρνηση ε, για ε, να εξετάσω ορισμένα οικονομικά στοιχεία συγκεκριμένων τομέων του δημοσίου. Και αυτά φαίνονται αναλυτικά στις απαντήσει μου στο ερωτηματολόγιο. Όσον αφορά ε, την, ε, την προσέγγιση μου ε, προς την Κοκομπού, πιστεύω ότι απαιτείται ο μέγιστος βαθμός συνεργασίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο ελεκτικό συνέδριο και στην Κοκομπού. Εάν διοριστώ, προτίθεμαι να παρουσιάζομαι ενώπιόν σας και επίσημα και ανεπίσημα. Δεν γνωρίζω ποιο τομέα αρμοδιότητας θα αναλάβω, θα μου αναφέσει ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνεδρίου, αλλά πιστεύω ότι αν πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο ενδιαφέρεστε κι εσείς και αισθάνεστε ότι πρέπει να μου τηλεφωνήσετε, να μου στείλετε ένα ε, email, τότε ε, θα σας δώσω, εάν θέλετε και εσείς βεβαίως, και τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική μου διεύθυνση για να μπορούμε να έχουμε στενή επαφή. Εάν θεωρούμε και αν θεωρείτε ότι προκύπτει ανάγκη. Πιστεύω ακράβαντα στη στενή σχέση ανάμεσα στους άμεσα εκλεγμένους που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των φορολογουμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ταυτόχρονα είναι σημαντικό ο, ο ρόλο και των μέλλον του Ελεκτικού Συνεδρίου γιατί εξασφαλίζουν ότι τα χρήματα αυτά σωστά. Θα, θα, ε, θα, θα προτείνω ε, την ενεργό συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε ε, έλεγχο. Θα προτείνω τη συμμετοχή στα αρχικά στάδια, στα στάδια σχεδιασμού, στις αποστολές και η εμπειρία μου, η επαγγελματική μου εμπειρία, νομίζω ότι θα προσδώσει προσθέμενη αξία. Εάν δηλαδή συμμετέχω και στο σχεδιασμό και στη διεξαγωγή και στην ολοκλήρωση των ελέγχων. Θα ήθελα λοιπόν να είμαι ε, ένα ε, μέλος του ελεκτικού συνεδρίου το οποίο ε, θα έχει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο. Προσωπική μου προσέγγιση είναι ένας τομέας στον οποίο έχω ιδιαίτερη εμπειρία. το value for money, την οικονομική αποδοτικότητα και, στην, και, στο, και, στον ιδιωτικό τομέα. Κάθε φορά έθετα το ερώτημα αυτό. Ε, θα είναι, είναι αποδοτική αυτή η δαπάνη. Αυτό λοιπόν ε, θέτω πάντα σε ερώτημα. Εγώ τα δικά μου χρήματα θα τα δαπανούσα προς την κατεύθυνση αυτή, θα περίμενα περισσότερα και θα έκανα τα πράγματα διαφορετικά την επόμενη φορά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η προσέγγιση που έχει άμεσο αντίκτυπο σε αυτό που προσδοκούν από εμάς και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να επεκταθώ λίγο περισσότερο στην ερώτηση παριθμών 4 που αναφέρεται στην απαλλαγή από τις προηγούμενες μου αρμοδιότητες ε, στα για τα καθήκοντα management. Έστειλα στην κυρία Αγιάλα, στην εισηγήτρια, μία σειρά επιστολών που επιβεβαιώνουν την παρέτησή μου από τις διάφορες θέσεις που κατήχα. και βεβαίω είμαι έτοιμο να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα τυχόν έχετε. Σα ευχαριστώ. Κυρία Γιάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω κύριε, κύριε Σύ. Σας ευχαριστώ και για τις επιστολές τι οποίε θα δώσω και στον κύριο Ντεματζίστρη, έτσι ώστε να πάρουν αντίγραφα όλοι οι συνάδελφοι, γιατί ήταν μία από τι ερωτήσει που θα σα έκανα. Α. Δεν ακούτε τη διερμηνία. Να σα επαναλάβω λοιπόν αυτά τα οποία είπα, σα καλωσορίζω στην Επιτροπή μας και επίση σας ε, ευχαριστώ και για το γεγονό ότι μου στείλατε αυτές τις επιστολές όπου φαίνεται η παρέτησή σα από όλα τα αξιώματά και από όλε τι θέσει. Γιατί έχετε ένα. Ε, ε είσαστε πολύ νέο, ε, σας προσωπικό σχόλιο βεβαίω, και έχετε τρομερή εμπειρία. Βεβαίω αυτό το είπα ε, εν παρενθέσει. Πραγματικά μακάρι όλοι να αξιοποιούσαν την νεαρή του ηλικία όπως την αξιοποιήσατε κι εσεί. Λοιπόν, ένα από τα προβλήματα είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν φαινόταν στι απαντήσεις σα η παρέτησή σα. από την ομάδα εξέταση συμφωνία Σαντάντριου και με εντυπωσίασε ε, αυτό το ζήτημα. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με την παρακολούθηση ε, της δαπάνης των χρημάτων ε, για, την, ε, για την εγκατάλειψη της τρομοκρατίας λοιπά, Όλα αυτά με εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα, πάντως μας απαντήσατε. Τώρα, δύο σημεία τα οποία μου προκαλούν ανησυχία. Και να δούμε τι θα μας απαντήσετε. Πρώτα απ' όλα, όταν έχουμε την, την ερώτηση ε, θα δημοσιεύατε τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Είστε ο μόνο που απαντά ναι αν το κάνουν όλα τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου. Οι υπόλοιποι δηλαδή είναι έτοιμοι να το πράξουν. Να δώσουν τη φορολογική δήλωση. Βεβαίω δίνετε τη φορολογική σας δήλωση στον πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου. Αλλά είναι παράδοση ε, στο κοινοβούλιο να ζητάμε εμεί να δημοσιεύονται αυτέ οι δηλώσει ε, συμφερόντων. Καταλαβαίνω ότι εσείς γνωρίζετε πολύ καλά το κώδικα δεντολογίας, απαντάτε με ιδιαίτερο επαγγελματισμό, θα θέλαμε όμω να είστε πιο σαφείς όσον αφορά την αποδοχή αυτή τη δημοσίευση. Δεύτερον, είσαστε ιδιαίτερα ειλικρινείς όταν στην ερώτηση 7, εκεί που σας ρωτάμε πώς αντιμετωπίζετε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας ή απάτης ή και δωροδοκίας, με ενεχόμενους από το κράτος μέλους καταγωγής σας, εσείς πολύ σαφώς λέτε ότι θα ζητούσατε από τον πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου να αναλάβει την υπόθεση αυτή ένα άλλο μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Γιατί, ε, πώς το βλέπετε το ζήτημα αυτό, μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα. Τώρα, κάτι άλλο. Όσον αφορά ε, τις, ε, τα προσόντα σα, ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια ε, κάπως διαφορετική απάντηση όσον αφορά τη χρησιμότητα ή μη των εθνικών δηλώσεων. Και επειδή είστε και επαγγελματία, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ζήτημα. Γιατί μερικέ φορέ μπορεί τελικά να καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για να πάρουμε αυτές τις δηλώσεις. Και εσείς δίνεται κάπως ε, μία διαφοροποιημένη απάντηση να αφορά το αν είναι χρήσιμες ή όχι. Και κάτι άλλο. Μου αρέσει αυτό, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό που αναφέρεται ε, ανάμεσα στον ελεκτή και τον ελεγχόμενο. Και εσείς λοιπόν, ε, πέραν το σχέσιο με το ελεκτικό συνέδριο, ε, θέτεται το ερώτημα, το, ζήτημα ότι μπορεί δηλαδή να, αντλήσουμε, στοιχεία από τον ελεγχόμενο. Δηλαδή ο ελεγχόμενος να μην θεωρεί τον εαυτό του θύμα αλλά ε, να, είναι, να συμμετέχει και να συνεργάζεται σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό νομίζω ότι είναι ουσιαστική σημασία. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό που το λέτε ω υποψήφιο. Και τέλο, όσον αφορά τα follow ups τα οποία ε, χρειαζόμαστε, πώ το βλέπετε το ζήτημα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το θέτουμε όταν, θέτ, όταν ε, ο στόχος μας είναι ο έλεγχος ποιότητας. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν τα follow-ups αυτά. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ για αυτές τις ερωτήσεις. Θα τις απαντήσω με τη σειρά που τις κάνατε. Πρώτα απ' όλα, για την ομάδα εξέτασης της συμφωνίας ε, του Σεντ Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα βοήθησαν πάρα πολύ την Ιρλανδία και ένας ε, τρόπος βοήθειας ήταν ε, οικονομική στήριξη στην ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία. Μου ζητήθηκε λοιπόν να εξετάσω ένα από τα εκτελεστικά όργανα της Συμφωνίας Μεγάλης Παρασκευής πριν από 10 χρόνια. Υπήρχε λοιπόν άλλη μια συμφωνία του Σεντ του 2006 και με βάση αυτή την συμφωνία μου ζητήθηκε να εξετάσω την αποτελεσματικότητα και βάσει χρηματικών όρων ε, κάποιων ε, θεσμικών οργάνων που ασχολούνταν με τουρισμό, υγεία και άλλους τομείς εξετάσαμε την διαχείριση αυτών των θεσμικών οργάνων, είχαμε δημόσιες συναντήσεις ε, και υποβάλαμε μία έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο Βορρά Νότου που αποτελείται βεβαίω από υπουργού από τον Βορρά και από τον Νότο. Σας έχω λοιπόν υποβάλει και ένα σημείωμα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιρλανδίας που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή μου και το ότι ολοκληρώθηκε η συμμετοχή μου. Αυτά ως προς αυτό. Τώρα, για το ερώτημα που αφορά τη δημοσίευση των συμφερόντων μου. Που δεν έχω κανένα πρόβλημα να δημοσιευτεί τώρα ή να το δώσω σε οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής ε, που θέλει ή να το δημοσιεύσω κι εγώ στο στην ιστοσελίδα του ελεγκτικού συνεδρίου. Ένα πρόβλημα. Δεν ήθελα να θέσω κανέναν όρο. Ευχαρίστως να σας διαβεβαιώσω πως είμαι διατεθειμένος να το δημοσιεύσω εάν το επιθυμείτε εσείς ή οποιοδήποτε μέλος επιτροπής. Όσον αφορά τυχόν παρατυπίες και απάτες. Υπάρχει μια οδηγία που αφορά το ελεγκτικό συνέδριο του 2004 και εγώ θα την ακολουθήσω πλήρως αν τύχει να υποπέσει στην αντίληψή μου κάποια απάτη είτε στη δική μου χώρα είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε οικονομική ύφεση στην Ευρώπη. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Πρέπει λοιπόν να είναι απολύτω σίγουροι πως οποιοδήποτε αναμειγνύεται τα ευρωπαϊκά οικονομικά θα είναι πολύ υπεύθυνο και θα αντιμετωπίσει πλήρως οποιασδήποτε υποψία απάτης. Η δηλώση που έκανα για την ε, τυχόν σύγκρουση συμφερόντων είναι το τι θα έκανα εγώ εάν υπήρχε τέτοια σύγκρουση συμφέροντων. Και βεβαίως προφανώς δεν θα μπορούσα να ελέγξω κάτι εάν υπήρχε τέτοια σύγκρουση συμφέροντων. Δεν νομίζω να υπάρχει, απλά θεώρησα καλό να αναφέρω το τι θα έκανα εάν προέκυπτε κάτι τέτοιο όσον αφορά δε τις εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Νομίζω πως είναι σημαντικές, εγώ είμαι υπέρ των δηλώσεων αυτών αυτή τη στιγμή μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο σημαντικούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ελεγκτή για να υπάρχει διαβεβαίωση για τα συστήματα ελέγχου και αν ο ελεγκτής είναι πιο σίγουρος για τα συστήματα ελέγχου που υπάρχουν, σημαίνει πως απαιτείται λιγότερος ουσιαστικός έλεγχος, κατά το οποίο βέβαια μπορεί να εξοικονομήσει κονδύλια και να ολοκληρωθεί ευκολό, γρηγορότερα ο έλεγχος και να επικεντρωθεί σε άλλους πιθανώς πιο ουσιαστικού τομείς ο ελεγκτής. Δεύτερον, οι εθνικές δηλώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, ως ε, ελεγκτικά τεκμήρια για να μειωθεί έτσι ουσιαστικός έλεγχος ο οποίος θα απαιτείται και άρα να γλιτώσουμε χρήματα. Αλλά εθνικές αυτές διαβεβαιώσεις αξίζουν βεβαίω μόνο όσο και ο έλεγχος που προηγήθηκε. Οπότε πρέπει να υπάρξει κάποια εναρμόνιση των ελεγκτικών προτύπων, γιατί σε διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικά συστήματα, άλλες εφαρμόζουν λογιστική εισόδων και άλλες όχι, άλλα μπορούν να ελέγξουν τους τελικούς δικαιούχους απευθείας και άλλα όχι, άλλες ε, κοιτούν και τον έλεγχο και τον εξωτερικό έλεγχο. Οπότε, για να υπάρξει ενιαία εφαρμογή και στα 27 κρατημέλη, θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα της πιλωτικής μελέτης για να δούμε το πώς, όχι το εάν, το πώς θα χρησιμοποιηθούν από το ελεγκτικό συνέδριο οι εθνικές ε, αυτές ε, διαβεβαιώσεις στο μέλλον. Δηλώσεις αξιοπιστίας. Σημειώνω αυτό το οποίο είπατε βεβαίως για το ότι ο ελεγχόμενος ε, συμμετέχει. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ πέρα πως σε τελική ανάλυση εξυπηρετούμε τους Ευρωπαίους φορολογούμενους και αυτούς οι οποίοι και αυτοί οι οποίοι ξοδεύουν τα λεφτά και αυτοί οι οποίοι κάνουν τη δήλωση πρέπει να αντιληφθούν πως ε, πρέπει να προσθέσουμε κάποια αξία και να δούμε ποιο όφελος θα έχουμε και του χρόνου και του παραχρόνου. Όσον αφορά τώρα το τι συνέχεια θα δοθεί σε έναν έλεγχο, ο έλεγχος είναι σοβαρή δουλειά, είναι ακριβή υπόθεση και είναι αναγκαίος. Αλλά για να μειωθεί αυτό το κόστος και να αυξηθεί το όφελος, Πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Δεν έχει νόημα να κάνουμε μια ερώτηση. Να κάνουμε μια σύσταση και του χρόνου να μην βλέπουμε τι έγινε με αυτές τις συστάσεις σε όλους τους ελέγχους, στους οποίους θα αναμειχθώ. Θα προσπαθήσω να δω εάν αντλήθηκαν διδάγματα από το παρελθόν και πώς εφαρμόζονται στο παρόν. Νομίζω απάντησα και τις πέντε ερωτήσεις. Αν ε, έχετε και άλλες, ευχαρίστω. Κύριε Μακοβέη. Τρεις ερωτήσεις, θα είμαι πολύ σύντομη. Πρώτη. Τι πιστεύετε για το σύστημα των ε, συγκεκριμένων, των ΤΑΣ εν πάση περιπτώσει. Πιστεύετε ότι πρέπει να τελειοποιηθεί το σύστημα αυτό ή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παραμείνει ως έχει. Σχετικά με την ε, σχέση αξίας και τιμήματος να αναφερθώ στις δημόσιες προμήθειες που είναι ο τομέας που είναι ο πλέον στη διαφθορά όπως επίσης και στα περιφερειακά ταμεία. Έχετε κάποια εμπειρία γύρω από αυτά. Είστε έτοιμος να εργαστείτε σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή διαφθορά στις δημόσιες προμήθειες που οδηγεί σε απάτες. Και τρίτη ερώτηση, το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να συνεργαστεί και με εσωτερικά αρμόδια όργανα. Υπάρχουν ορισμένα ελεγκτικά συνέδρια στα κράτη-μέλη που δεν είναι πολύ διαθέσιμα για συνεργασία και δεν είναι διατεθειμένα να εργαστούν για διάφορους λόγους με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Είστε προετοιμασμένος γι' αυτό, τι σκοπεύετε να κάνετε, ποια είναι η στρατηγική σας. Θα ήμουν υπέρ της διαδικασίας η οποία ακολουθείται σχετικά με τις δηλώσεις αξιοπιστίας. Καταρχάς συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στα θέματα των ελέγχων. Εγώ λέω ότι είναι προτιμότερο να μάθεις κάποιον ε, να ψαρεύει μόνος του παρά να του κάνεις δώρο ένα ψάρι για να τραφεί για μια συγκεκριμένη μέρα. Εδώ είναι και το ενδιαφέρον των ελέγχων. Να ενθαρρύνει κανείς ένα οργανισμό να ασκεί ελέγχους σε συνεχή βάση. Έτσι δεν λειτουργείς σαν ένας ορκωτός ελεγχτής ο οποίος εκ των υστέρων βλέπεις το τι έχει γίνει, αλλά σαν κάποιος ο οποίος σε μόνιμη βάση προωθεί την κουλτούρα της, της κανονικότητας αν θέλετε και του ελέγχου. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ελέγχου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα και είναι απαραίτητο να διανυθεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επιθυμητό επίπεδο συμβατότητα σε 95%. Νομίζω ότι αυτή η αντιμετώπιση σαφώς και μεγιστοποιεί την προστιθέμενη αξία της ε, διαδικασίας ελέγχου και ελαχιστοποιεί το κόστος που απαιτείται για να φτάσει κανείς σε αυτή τη φάση. Θα είμαι λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικός σε οποιαδήποτε μορφή ελέγχου συμμετέχω, έτσι ώστε η διαδικασία αξιολόγησης του περιβάλλοντος ελέγχου να έχει προηγηθεί, να είναι προσεκτική και να έχουν υπάρξει και δοκιμαστικές ε, περίοδοι των μορφών αυτών ελέγχου, σαν παράδειγμα τα δείγματα τα οποία έχουν συγκεντρωθεί η δειγματοληψία να αντιπροσωπεύει ένα ομοιογενές πεδίο ενδιαφερομένων εμπλεκομένων. Όταν δει κανείς την διαδικασία η οποία περιέχεται σε μία δήλωση τέτοιου είδους αξιοπιστίας είναι κάτι το ιδιαίτερα περίπλοκο. Και η δυνατότητα την οποία παρουσιάζει μια τέτοια ε, δήλωση είναι κάτι το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί από την Επιτροπή σας και από τον Ευρωπαίο πολίτη. Σχετικά τώρα με το κόστος και το όφελος. Οι δημόσιες προμήθειες έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. 120 δις δαπανώνται ε, σε επίπεδο κοινοτικού προϋπολογισμού, το 1 τρίτο πηγαίνει στη συνοχή, το 85% πηγαίνει σε άλλες δαπάνες και ένα μικρότερο ποσοστό ε, περνάει μέσα από τα κοινοτικά όργανα. Οι έλεγχοι θα πρέπει λοιπόν να γίνονται, οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι διαφανείς, ε, θα πρέπει να προσφέρονται σε εξωτερικές και εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου. όσοι είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση του δημοσίου χρήματος ε, είναι απαραίτητο να γίνεται ο έλεγχος γιατί αν δεν γίνεται τότε ε, στην ουσία υπάρχει μια διαδικασία προδοσίας της εμπιστοσύνης του Ευρωπαίου πολίτη. Αυτό είναι ευθύνη κάθε μέλους του ελεγκτικού συνεδρίου ο οποίος θα πρέπει να προχωρήσει στο να γίνεται αυτό το οποίο, για το οποίο έχει τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη θέση. Οι δημόσιες προμήθειες λοιπόν είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας γιατί ο κόσμος δαπανά τα χρήματά του και πρέπει να γνωρίζει και μέσω των δηλώσεων αξιοπιστίας ότι δεν πηγαίνουν χαμένα τα χρήματα, τα χρήματα αυτά σχετικά τώρα με τα εθνικά συστήματα ε, ελέγχου και ελεγκτικά σώματα. Το ίδιο κάνουμε εμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Ελέγχουμε τις δαπάνες, είμαστε ένα είδος εξωτερικών ελεγκτών Και αν τα σώματα αυτά δεν είναι διατευστούν σε διάφορους τομείς υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Καταρχάς, κάποιος που δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μου θα έρθω σε επαφή προσωπική μαζί του, θα του ζητήσω τους λόγους και τις εξηγήσει. Είμαι λογικός άνθρωπος και θα προσπαθήσω να τους πείσω ότι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν και ότι αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να ολοκληρωθεί και είναι μια διαδικασία που προσθέτει αξία στον έλεγχο. Εδώ και λίγα χρόνια θα φανταζόμουν ότι ε, οι Ευρωπαίοι ελεγκτές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είχαν μια ξεκάθαρη, ε, ξεκάθαρα αρνητική σχέση γιατί είχαμε αρνητικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει ακόμα και σε τομείς όπως η Γεωργία. Και διάβασα τα πρακτικά της ακρόασης ε, του κυρίου Σεμέτα, του αρμοδίου που είναι υπεύθυνο για τις ελεγκτικές διαδικασίες και είπε ότι η θετική τάση είναι βασική του προτεραιότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι η αναφορά περιπτώσεων το να είναι κανείς αναφερόμενος στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου όλο και λιγότερο από χρόνο σε χρόνο, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ελκυστικό και για τα αντίστοιχα κράτη-μέλη. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει μια θετική σχέση ε, του ελεγκτικού συνεδρίου με τα εθνικά ελεγκτικά σώματα και όταν υπάρχουν αρνητικές αντιδράσεις θα προσπαθήσω να τις αντιμετωπίσω με θετικό πνεύμα. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω αν έχετε συμπληρωματικές. Ένα μικρό σχόλιο. Θα βρείτε στα κράτη-μέλη, σε κάποια κράτη-μέλη, σώματα τα οποία δεν θέλουν να συνεργαστούν, όχι ότι δεν μπορούν. Το θέμα δεν είναι να τους πείσετε, αλλά είναι τμήμα ενός συστήματος το οποίο προστατεύει α, τις παρατυπίες. Πρέπει να είστε απόλυτα διαθέσιμος γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές σας και προφανώς θα τις λάβω υπόψη. Ο δημοσιονομικός κανονισμός γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκ νέου και αν πάρω τη συγκεκριμένη θέση θα έχω ίσως τη δυνατότητα να αντιμετωπίσω συγκεκριμένα παραδείγματα αυτού το οποίο λέτε έτσι ώστε να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε το δημοσιονομικό κανονισμό όπου χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω την άποψή σας όσον αφορά την ποιότητα του λογιστικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα. Διότι οι πολίτες και οι πρόσωποι των πολιτών, ε, προκειμένου τα μέλη του Κοινοβουλίου, μπορούν να αναρωτηθούν μετά από τα γεγονότα στην Ελλάδα για την ποιότητα ε, των ε, ε, εθνικών αυτών εκθέσεων και την ποιότητα του ελέγχου και νομίζω εξάλλου ότι αν αναρωτηθούμε για την ποιότητα αυτών των στοιχείων και στα άλλα κράτη-μέλη που τοποθετήθηκαν για το θέμα της Ελλάδας, βλέπουμε ότι τέτοιες λογιστικές ακροβασίες γίνονται και σε άλλα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν κανείς δεν έχει το δικαίωμα να δώσει διδάγματα στους υπολείπους. Όσον αφορά το ελεκτικό συνέδριο, επειδή εάν ε, διοριστείτε θα, θα ασκήσετε έλεγχο, εσείς θα δεχόσασταν να είσαστε ο ίδιος ελεγχόμενος ε, την κατάλληλη στιγμή στα πλαίσια του peer review. Και, ποιος, και ποια ε, είναι η άποψή σας για το ζήτημα αυτό. Και για, τις, και το ελεκτικό έργο του ελεκτικού συνεδρίου στο σύνολό του. Απάντηση. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όσον αφορά την ποιότητα του ελέγχου στα δημόσια τομέα, θα ήθελα να κάνω την εξή παρατήρηση. Το value for money δεν αναφέρεται στη συνθήκη. Όμως, το ελεκτικό συνέδριο αναλαμβάνει αυτούς τους ελέγχους επιδόσεων ε, και αυτές τις ειδικέ εκθέσεις. Ένα από τα ζητήματα που αφορούν τις ειδικέ εκθέσεις και παρατήρησα εγώ είναι ότι χρειάζονται 26 μήνες από την πρώτη ε, πρόταση για μια διέκριση μέχρι τη δημοσίευση. Νομίζω λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε επιτάχυση των διαδικασιών. Γιατί? Ε, ο λόγο για τον οποίο ε, υπάρχει ανάγκη αυτέ τι εκθέσει είναι πολύ συγκεκριμένο. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να περνάει τόσο χρόνο ε, και να περιμένουν οι πολίτε τόσο χρόνο μέχρι να πάρουν απάντηση πρέπει να δουν την απάντηση στα ζητήματα τα οποία θίγονται στην ειδική έκθεση. Άρα λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο τομέα, ε, ο δημόσιο τομέα είναι μάλλον διαφορετικό ε, σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και άρα θα έλεγα ότι και ποιότητα αλλά και ταχύτητα. Γιατί βεβαίως ε, καταλαβαίνετε ότι κανείς ε, ζυγίζει τα δύο στοιχεία. Από τη μια ε, είναι σημαντικό το να έχει κανείς πληροφορίες εδώ και τώρα ε, και που πολλές φορές αυτή είναι η ορθή προσέγγιση, αλλά από την άλλη παίρνει πιο πλήρες πληροφορίες αν κανείς περιμένει λίγο χρονικό διάστημα. Επίσης, αναφέρθηκε ένα ζήτημα σε σχέση με ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Δεν είμαι μέλος του ηλεκτρικού συνεδρίου τώρα και η μόνη μου ενημέρωση προέρχεται από τον τύπο και τις εφημερίδες. Όμως, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο αναφέρθηκε σε γενικότερο επίπεδο ε, για ε, την δημιουργική λογιστική. Και μπορώ να σας πω την προσωπική μου άποψη για το ζήτημα αυτό. Ως ε, πολίτης και ως επαγγελματίας, ως ορκωτής λογιστής, ότι εμείς απαιτούμε συνέπεια και η λογιστική πρέπει να είναι η ίδια και πέρυσι και φέτος και του χρόνου. Και σε δύο χρόνια. Γιατί διαφορετικά, αν δεν υπάρχει συνέπεια, οι πληροφορίες ε, που αφορούν τους λογαριασμούς δεν έχουν κανένα νόημα. Άρα λοιπόν συνέπεια. Είναι πολύ σημαντική η αρχή αυτή της συνέπειας. Και αν κάποιος αλλάζει την πολιτιστική του στον τομέα της λογιστικής, τότε πρέπει να ε, αναφέρει και τα, ε, και τα στοιχεία με την, ε, τα προηγούμενα και να τα συγκρίνει με τα νέα στοιχεία τα οποία προέρχονται από την αλλαγή πολιτική στον τομέα τη λογιστική. Για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι λογιστικέ ακροβασίε, πρέπει να είμαστε καλοί λογιστέ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πρέπει να μπορούμε να, να βλέπουμε παντού και να αποκαλύπτουμε τις απάτες. Αν κανείς δημιουργήσει τη φήμη ότι αποκαλύπτει τι απάτε. Αν κανείς αποκτήσει τη φήμη ότι γνωρίζει τα λογιστικά, τότε δεν πρόκειται κανείς, δεν πρόκειται οι υπόλοιποι να δοκιμάζουν τέτοια παιχνίδια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το ελεκτικό συνέδριο έχει καλή φήμη και πρέπει να προστατεύσει αυτή την καλή φήμη του. Και να μην επιτρέπει από τους υπόλοιπους να ε, του δημιουργούν αυτά τα προβλήματα ε, αλλάζοντας τα στοιχεία ή αλλάζοντας τη βάση με την οποία ε, προκύπτουν τα στοιχεία αυτά. Δεν μπορεί κανείς να αλλάζει τα στατιστικά επειδή ακριβώς αλλάζει το άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για τα στατιστικά αυτά τα στοιχεία. Εάν το, τώρα, όσον αφορά τον έλεγχο των μελών του ελεκτικού συνεδρίου, βεβαίω πρέπει και εμεί να υφιστάμεθα σε έλεγχο. Ε, κάθε χρόνο γίνεται αυτό από ανεξάρτητους ε, ε, λογιστές που προβαίνουν σε ανάλυση αξιοπιστίας, ανάλυση δηλώσεων αξιοπιστίας και ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται peer review, έλεγχος ομοτήμων. Δεν έχει γίνει κάτι τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά φυσικά θα πρέπει και εμεί να εξετάζουμε τον εαυτό μα. Θα ήταν ιδιαίτερα εγωιστικό εκ μέρου του Ελεκτικού Συνεδρίου να επιμένει ε, στον έλεγχο όλων των υπολείπων, αλλά να μην μπορεί να δεχθεί τον έλεγχο, ε, ε, τον έλεγχο το ίδιο το ελεκτικό συνέδριο, γιατί όλα αυτά είναι μέρος μιας διαφανούς και δίκαιας πολιτικής. Ευχαριστώ, Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Πράγματι μας κάνετε καλή εντύπωση, χαιρόμαστε που σας ακούμε και ελπίζω πράγματι αυτή η χαρά να παραμείνει και στην υπόλοιπη συνεργασία μας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο είπατε. Ξέρετε, για μας είναι ζήτημα άξιο πιστείας του να μην προστατεύουν τις δικές τους χώρες τα μέλη του Ελληνικού Συνεδρίου, γιατί ακούγονται διάφορα, γιατί άρα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες είναι οι πιέσεις και οι επιρροές. Ξέρουμε βέβαια πως δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ε, εάν θα έρχεστε ε, εδώ πέρα. Θα ήθελα, δεν υπάρχει ερώτηση, να σας παρακαλέσω να, έρκε, να έρχεστε γιατί είναι δύσκολες οι επικοινωνίες με το Λουξεμβούργο και αυτό είναι πρόβλημα και για τη συνεργασία που νομίζω ότι μπορεί να είναι καλύτερη. Εάν π.χ. οι ειδικέ εκθέσεις έρχονται πιο σύντομα, έχουν μικρότερες ε, προθεσμίες ε, και είναι πιο ισορροπημένες ε, και είναι πιο ουσιαστικέ, νομίζω θα είναι καλύτερο αυτό και το είπα και σε κάποιου υποψηφίου. Η δική μου η κριτική είναι πω θέλουμε περισσότερη βοήθεια από το συνέδριο, χρειαζόμαστε περισσότερα θέματα και να υπάρχει και μια πρόβλεψη Γιατί λαμβάνουμε κάποιε πληροφορίε και ορισμένε φορέ πρέπει να δούμε μόνοι μα τα κάνουμε. Γιατί είναι το θέμα και του προσωπικού και τη αποκέντρωση της, ε, ε, του ότι αναθε, ανατίθενται δουλειές σε εξωτερικούς συνεργάτες εδώ και χρόνια και δεν είχαμε κάποιο σχετικό έγγραφο όσον αφορά την ε, γενικότερη πολιτική. Το ίδιο ισχύει και για την ύπατη εκπρόσωπο που έχει κάνει το γύρο του κόσμου και αναρωτιόμαστε τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν θέλω βέβαιω να σας δυσκολέψω την δουλειά ενώ δεν ξεκινήσατε ακόμα. Απλά σας αναφέρω πώς έχουν τα, τα πράγματα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γκρέσλε για τις ερωτήσεις. Βεβαίως να βασιστείτε σε αυτά τα οποία είπα. Οπότε έρχομαι στις Βρυξέλλες, θα ενημερώνω την Επιτροπή, γιατί όσο περισσότερη δημοκρατία υπάρχει, και όσο περισσότερο είστε εσείς ενημεροί ή τόσο το καλύτερο το όφελος για το φορολογούμενο. Είχα κάποιες ε, συζητήσεις με λίγους από εσάς και ο ενθουσιασμός για την δουλειά σας είναι εξαιρετικός και χαίρομαι. Και ειδικά όταν διαλέγουμε θέματα για τις ειδικέ εκθέσεις πρέπει να λάβουμε υπόψη της Απόψης της Επιτροπής σας γιατί βεβαίως όταν λέμε ότι θα κάνουμε μια τέτοια έκθεση ε, κάτι τέτοιο έχει αμέσως θετικά αποτελέσματα μεταξύ των, των ελεγχομένων και καθώς ε, οι επιτροπές αυτές ε, ασχολούνται περισσότερο με την αποδοτικότητα του κεφαλαίου, είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Όσον αφορά την εθνική και την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα για τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου και οποιοδήποτε άλλου ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου. Πρέπει να τονίσω πως εάν μου δώσετε βεβαίω αυτή τη θέση θα είμαι υπάλληλο ε, των ε, πολιτών της Ευρώπης. Και υπ' αυτή την, ε, την ιδιότητα θα θυμώ βεβαίω πως ο εργοδότης μου είναι οι λαοί της Ευρώπης. Και εγώ θα βοηθήσω και θα με βοηθήσουν κυρίως βεβαίω τα μέλη της, ε, της Επιτροπής σας, γιατί σε εσά έχει ανατεθεί από τους πολίτες της Ευρώπης να έρθετε σε επαφή μαζί μας για να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο τα κονδύλια που έχουν εμπιστευτεί στη διαχείρισή μας οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Νομίζω πως ε, απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Αν όχι, παρακαλώ πείτε μου, κύριε Γκρέσλε. Ναι, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ίσως δεν παρακολούθησα πάρα πολύ καλά την παρουσίαση, την απάντηση μάλλον, αλλά αν κατάλαβα καλά, ε, είπατε ότι θα σας βοηθήσουμε. Η συνάδελφός μου το αντίθετο ζητούσε, εσείς να μας βοηθήσετε. Μπας περιπτώσει αυτό δεν είναι, ε, είναι δευτερεύον. Ένα τελικό σημείο το οποίο είναι θετικό. Όλος ο ενθουσιασμός τον οποίο επιδεικνύεται για τα επόμενα δύο χρόνια είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. η διάρκεια της περίοδου είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχω εγώ. Αν μετά από μια χρονική περίοδο θεωρήσετε ότι έχω κάνει καλή δουλειά, να μου το πείτε, να το πείτε και στην κυβέρνησή μου. Ευχαριστώ κυρία Αγιάλα Σέντερ. Σας ευχαριστούμε όλους. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9.